Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη συνεδρίαση. Ε, σας καλημερίζω όλου και ξεκινάμε με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έγκριση τη ημερήσια διάταξη, και να κάνω μια ανακοίνωση. Ε, το σημείο 18, η έκθεση Ρώση δηλαδή, θα είναι το πρώτο θέμα αύριο το απόγευμα. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη υπό τη μορφή αυτή και προχωράμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσια διάταξη. Ε, το, το γλωσσικό καθεστώς ε, είναι πλήρες εκτός από εστονικά. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εστονικά. Ε, επίσης, μία ανακοίνωση για την ε, οδηγία για την ε, ποιότητα των καυσίμων ε, και τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Δεν υπήρξε πλειοψηφία. Ψήφισαν 89 υπέρ, 128 κατά και 128 αποχές. Ε, είμαστε λοιπόν περίεργοι τι θα προτείνει η Κομισιόν. Αύριο το Αύριο το πρωί θα έχουμε εδώ μια ε, ομάδα από το κανάλι VDR της Γερμανίας και στις 8 Μαρτίου θα ε, οργανώσουμε ένα σεμινάριο στις 9.30 στην αίθουσα aspg 3 Και ε, ένα ακόμα σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 20, στις 20 Μαρτίου 10 η ώρα, SP3G3 ε, είναι η αίθουσα ε, και έχει να κάνει με ε, ένα ευρωπαϊκό σύστημα τελών. Έκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 19ης-20ης δεκεμβριου Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται λοιπόν. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης ε, και την έκθεση του Καρλ Σλούτερ. Έχουμε σήμερα ε, αρκετές ε, εκθέσεις στην ημερήσια διάταξη, όλες έχουν να κάνουν με την αλληλεία και η έκθεση του Καρλ Σλούτερ έχει να κάνει με το πολιτές σχέδιο για το απόθεμα Σολομού της Βαλτικής και την αλληλευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος. Του δίνω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σήμερα σου ειδικά. Eh, Ο Σολομός έχει μια ιστορία. Όταν ξεκίνησε η βιομηχανοποίηση στην ε, χώρα μου ε, στα μέσα της, ε, του 19ου αιώνα, στο, στη Σύμβαση των Εργαζομένων έλεγε ότι δεν επιτρεπόταν να τρώνε σολομό πάνω από έξι μέρες τη βδομάδα. Ήταν τόσο υψηλός αρχικός πληθυσμός που ε, ο Σολομός ήταν ε, το πιο φθηνό Σήμερα η κατάσταση είναι ε, διαφορετική. Οι περισσότεροι, στους περισσότερους ποταμούς της Βαλτικής οι Σολομοί απειλούνται ή έχουν εξαφανιστεί και το 90% του άγριου σολομού ε, στην, ε, γεννιέται στην, ε, σε δύο ποταμούς μόνο στην Βόρεια Σουηδία και Φιλανδία. Αυτοί οι δύο ποταμοί λοιπόν είναι η βάση για το συνολικό απόθεμα του άγριου σολομού. Και πέρα από την ε, καταστροφή του περιβάλλοντος ε, και ασθένειες έχουμε ε, χτίσει και πολλές εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικές οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα αλλά σημαίνει επίσης ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται οι σολό με τον ίδιο τρόπο στους ποταμούς. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι λόγοι που έχει μειωθεί το ε, το άγριο απόθεμα και έχουμε ε, επιβάλει τώρα ε, σε αυτούς, στους ιδιοκτήτες της εκεί να, να δημιουργήσουν νέα αποθέματα. Ε, τα οποία όμως ε, είναι νέα είδη, ε, τα οποία μεγαλώνουν γρήγορα, τα οποία όμως δεν είναι απαραίτητα εξίσου δυνατά. Τώρα λοιπόν αλλιεύουμε σολομό στην ανοιχτή θάλασσα, όπου αναμειγνύεται ο ο άγριος σολομός με τον ε, καλλιεργημένο σολομό και ο ε, ε, καλλιεργημένος συχνά δυσκολεύεται να επιστρέψει στα, αρχικά ύδατα. Ο άγριος σολομός λοιπόν έχει... Ο άγριος είναι πολύ πιο δυνατό είδος και... δεν ξέρουμε αν η σολομή που αλλιεύουμε είναι από τους αρχικούς ε, ε, από τους αρχικούς άγριους πληθυσμούς ή αν είναι ε, σολομή εκτροφής. Και γι' αυτό στην... στην έκθεσή μου προτείνω, στο σχέδιο γνωμοδότησης προτείνω να σταματήσουμε την αλληλεία του Σολομού στην ανοιχτή θάλασσα. Όταν λοιπόν εκτρέφουμε Σολομό στη Βαλτική, και ε, τον απελευθερώνουμε σε έναν ποταμό και κατόπιν ε, ε, έχουμε τα σκάφη στη Βαλτική που αλλιεύουν αυτά τα ψάρια. Είναι πολύ κακός τρόπος να πιάνει κανείς έτσι σολομούς εκτροφής. Εάν οι σολομοί αλλιεύονται κοντά στους ποταμούς όπου ε, γεννιούνται έτσι είναι ε, δυνατόν να αποφεύγουμε την αλληλεία ε, απειλούμενων αποθεμάτων. Η πρότασή μου λοιπόν είναι και έχω εισάγει μια μακρά μεταβατική περίοδο, διότι καταλαβαίνω ότι αν μειώσουμε την αλληλεία αυτό θα πλήξει διάφορα κράτη-μέλη με διαφορετικούς τρόπους, αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ε, για να αποκατασταθεί ο άγριο σολομό, ο οποίο είναι και το πιο ισχυρό είδο. Και ε, στις περιπτώσεις ε, όπου απελευθερώνει κανεί σε σολομούς εκτροφή, σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσει κανεί ένα είδο το οποίο γενετικά να μοιάζει τόσο πιο, όσο γίνεται πιο πολύ στο είδος που υπάρχει στον ποταμό στον οποίο απελευθερώνεται ο πληθυσμό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε λίγα να γίνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ε, αυτό είναι το βασικό στοιχείο της γνωμοδότησής μου. Άλλο ε, στοιχείο είναι να βελτιωθεί η ε, η λογοδοσία, η υποβολή εκθέσεων, διότι περίπου το μισό των Σολομών που αλλιεύονται σήμερα δεν, δεν αναφέρονται Και επίσης ε, στην αλληλεία αναψυχής ε, είναι Πολύτιμο ο κάθε σολομός ε, που αλλιεύεται. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη, καλύτερο έλεγχο των ε, ε, ψαριών αυτών που αλλιεύονται και θέλουμε μείωση αυτών των ψαριών από το, την εθνική ποσοστόση ώστε να έχουμε καλύτερη συνολική εικόνα των ψαριών που αλλιεύονται. Πάντως ε, η βασική ιδέα το να απελευθερώνουμε ε, σολομό εκτροφής για να τον αλλιεύσουμε κατόπιν ε, στις θάλασσες είναι ουσιαστικά σπατάλη χρημάτων και συνεπάγεται και την αλληλεία απειλούμενων αλλιών, σολομών που κατά τα άλλα θα είχαν δυνατότητες αποκατάστασης. Ευχαριστώ Κάλ Σλίτερ, ο Κρίστοφερ Φιέλνερ. Äh, e Και η Άννα Ρόσπαχ από το ECR. Αυτός είναι ο κατάλογος των ομιλητών, ο Κρίστοφερ Φιέλνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, καλούς Λίτερ. Καταρχήν ε, το θέμα ε, απαγόρευσης ε, της αλίας Σολομού στην ανοιχτή θάλασσα. Θα ήθελα να το εξετάσω αυτό εις βάθος, διότι όπως ε, είπες πρόκειται για μακροπρόθεσμα μέτρα και είναι πολύ πιθανό να είναι αυτό το μόνο, το μόνο δυνατό μέτρο, το μόνο πραγματοποιήσιμο μέτρο, ε, αλλά ε, έχω μια αίσθηση ότι η πρόκληση στην Αλία Σολομού είναι ότι είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στα διάφορα μέρη, διότι όπως είπες Καρλ, μιλάμε για πολύ διαφορετικούς πληθυσμούς γενετικά. Για παράδειγμα, στον κόλπο της Ρήγα υπάρχει ε, ένα απόθεμα Σόλομου και μήπως ε, είναι καλύτερο να έχουμε ένα σχέδιο αποκατάστασης ε, για κάθε πληθυσμό αντί να έχουμε ε, την ίδια ρύθμιση για όλους. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι κατά πόσο η απαγόρευση αλίας στην Βαλτική θα πρέπει να, αποτε... να καλύπτει όλη τη Βαλτική. Επιπλέον, Πιστεύω ότι έχει απόλυτα δίκιο όσον αφορά την, ε, την αρρύθμιστη αλία, αυτήν που δεν αναφέρεται. σε σχέση με άλλα ψάρια ανατόνο ε, ε, ο Σολομός ε, που, που αλλιεύεται για λόγους αναψυχής είναι πολύτιμος. Ε, μιλάμε όμως επίσης ε, για μεγάλο ποσοστό. Το ότι έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό μη αναφερόμενης αλληλείας, ε, μη καταχωρημένης αλληλείας έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Σολομός είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των αλληλεών που αλλιεύουν για αναψυχή. Ε, μπορεί όμως να διαπιστώσουμε ότι ακριβώς η ε, να να αποτελεί μέρος ε, του προβλήματος, γιατί αυτό εξαρτάται από ε, το ποια αποθέματα αλλιεύουν και πόσο ευαίσθητα είναι αυτά τα αποθέματα. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να έχουμε περισσότερα διαφορετικά προγράμματα και όχι ένα που να καλύπτει όλη τη Βαλτική. Αλλά θα το εξετάσω αυτό εις βάθος και θα επανέλθω, ιδιαίτερα στο θέμα της αλίας αναψυχής. Ευχαριστώ, Κρίστοφερ Φιέλνερ. Ο κύριος Παλάκης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να επιδοκιμάσω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολίτες πλαίσιο ε, και σχέδιο για το Σολομό της Βαλτικής και τους αλλοίς που στην περιοχή. Με το σχέδιο αυτοδράσης θα ε, αλλάξουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά της αλληλείας και θα επιτρέψουμε τη βιώσιμη διαχείριση των ελευτικών αποθεμάτων, διαφυλάσσοντας τη γενετική τους ε, ακαιρεότητα και την ε, βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ τον κύριο Σλίτερ για τις τροπολογίες του. Συμφωνώ με τις περισσότερες από αυτές, αλλά έχω και εγώ κάποιες επιφυλάξεις για την πρόταση σταδιακής κατάργησης ε, της αλίας ολομού στην ανοιχτή θάλασσα. Γιατί μια τέτοια απαγόρευση θα επηρεάσει ε, πολύ αρνητικά του αλεί σε συγκεκριμένε χώρε, ιδιαίτερα τη Βαλτική. Γι' αυτό και θα καταθέσω τροπολογία που θα λέω ότι η οικολογική ανάκαμψη του Σολομού και οι περιβαλλοντικέ ε, ανάγκε θα πρέπει να αντισταθμίσουν τα οικονομικά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να θεσπιστούν κάποια μέτρα διαχείριση ώστε να, συνεχίσει η αλία της Βαλτικής ε, και η αλία Σολομού της Βαλτικής να εξασφαλίζει θέσεις απασχόλησης και στο μέλλον. Η μείωση της ε, αλίας στην περιοχή της αλληλευτικής προσπάθειας θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης ε, με τους αλίες προκειμένου να έχουμε καλύτερη εφαρμογή αυτής της μείωσης της αλληλευτικής προσπάθειας και να εξασφαλίσουμε πραγματικά βιώσιμη αλληλεία, θα πρέπει να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο για τους φιλελεύθερους, ε, η, η συνάδελφος Μάνερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την ε, εξαιρετική, σαφέστατη και περιστατωμένη παρουσίαση που μας έκανε. Όπως ξέρουμε, στη Βαλτική θάλασσα τα αποθέματα άγριου σολομού βρίσκονται σε ενισχυτικά επίπεδα πια. Μα το λέει αυτό και ο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, αλλά και το Συμβούλιο τη Βαλτική Θάλασσα ε, θορυβήθηκε για την κατάσταση των αποθεμάτων άγριου σολομού. Αλλά και ε, τα ηχθίδια σολομού έχουν μειωθεί, οι νεαροί σολομοί έχουν μειωθεί, έχει αποδειχθεί αυτό και επιστημονικά, κάτι που θα επηρεάσει την μελλοντική ανασύσταση των πληθυσμών του Άγριου Σολομού είναι ένα σαφέ μήνυμα ότι η πολιτική τη Βαλτική θάλασσα ήταν αναποτελεσματική τα τελευταία χρόνια. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κάποια νέα μέτρα. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι ευπρόσδεκτη, είναι αξιόλογη. Χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση τη Ελία Σολομού για να διαφυλάξουμε τα αποθέματα αυτού του είδου. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Εξαιρετική η έκθεση του, η του μάλλον. Προτείνει ε, να είναι ακόμη πιο φιλόδοξη η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που είναι ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας και για τη συζήτησή μας. Ε, η μεικτή αλία είναι πολύ προβληματική στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί οι διάφορες λεκάνες απορροής μόνα δεν ε, μπορούν να διαχωριστούν. Και η μεικτή αλία δεν μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την προέλευση των ψαριών κάτι που αποβαίνει βάρος ουσιαστικά συγκεκριμένων ε, αλληλευτικών πληθυσμών, αλληλευτικών αποθεμάτων. Και μάλιστα στα δέλτα των ποταμών ε, καλό θα ήταν να επικεντρώνεται η αλληλεία και να μην ε, ε γίνεται μεικτή αλλήλευση στην ανοιχτή θάλασσα. ο περιορισμό αλληλεία στην ανοιχτή θάλασσα είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε την ανασύσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων. Αλλά φυσικά χρειαζόμαστε μεταβατικές περιόδους γι' αυτό, σταδιακή κατάργηση και όχι ο, ολοσχερή και ευνίδια, για να αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες. Κατά τη γνώμη μου, το πιο προβληματικό τμήμα της ε, γνωμοδότησης αφορά την ε, συγκεκριμένη περιοχή αλίευσης ε, του Σολομού. Γιατί λέμε ότι θα πρέπει να αλλιεύεται ο Σολομός ε, όταν αρχίζει και μπαίνει προς το ποτάμι όπου θα αναπαραχθεί. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το προσδιορίσουμε. Πάντως συμφωνώ και με τις τροπολογίες του εισηγητού που θεωρώ ότι ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Για, τους, ε, για την πολιτική ομάδα ECR, Άννα Ρόσπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Αγγλικά θα τα πω. Από μια ε, περιοχή, από μια χώρα της Βαλτικής που ασχολείται με την αλληλεία και με ανησυχεί η κατάσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων και οι μελλοντικές ε, αλληλευτικές προοπτικές. Δεν θέλουμε να χάσουμε την ευκαιρία αλλιεύση όλων στη Βαλτική θάλασσα, γιατί έτσι θα εξολοθρέψουμε τι αλλιευτικές μα κοινότητε. Δεν συμφωνώ με τον εισηγητή. Πολλέ χώρε γύρω από τη Βαλτική θάλασσα είναι αδύνατον να, να σταματήσουν την αλία τους στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν συμφωνώ με την κατάργηση, έστω και τη σταδιακή κατάργηση της αλίας στην ανοιχτή θάλασσα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η αλήφεις σολομών όταν βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής και όταν έχουν ε, ακόμη ε, αυγά. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η, παραγωγή, η αλίευση ολομού σε τέτοια φάση αναπαραγωγής. Συμφωνώ με τον εισηγητή για την μη δηλωμένη αλία. Η αδήλωτη αλία είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα δήλωσης και καταχώρησης. Επίσης, η ανακριβής δήλωση των αλίευμάτων υπάρχει κίνδυνο εδώ υπονόμευση των προσπαθειών που κάνουμε με την εφαρμογή των ποσοστώσεων για να διαφυλάξουμε τα αποθέματα. Σε ό,τι αφορά την ερασιτεχνική ελεία, η μία εμπορική ελεία θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτή στο συνυπολογισμό. Συμφωνώ με, πολλά στοιχεία της έκθεσης ε, Σλότερ, αλλά διαφωνώ με την ε, πρόταση για απαγόρευση της αλίας ε, Σολομού στην ανοιχτή θάλασσα, στη Βαλτική. Ευχαριστώ την Αναρόσπαχ και δίνω τώρα το λόγο στη Σάτου Χάση, παρακαλώ. Puheenjohtaja, ja ε, kiitoksia Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καρλ Σλότερ για την ε, θαυμάσια γνωμοδότησή του. Είναι πολύ εύστοχο το σχόλιο του ότι Η αλία Σολομών καλλιέργεια στην ανοιχτή θάλασσα είναι μια πραγματικά μάταιη και αναποτελεσματική αλία. Ε, επίσης δεν υπάρχει ένα κοινό ελευτικό απόθεμα Σολομού. Κάθε ποταμός έχει το δικό του ελευτικό απόθεμα με τα συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα βιολογικό γεγονός αυτή η ποικιλομορφία των γενετικών χαρακτηριστικών των Σολομών σε κάθε ποτάμι. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να προστατεύουμε τους ιδιαίτερους πληθυσμούς κάθε ποταμού. Και νομίζω ότι ο πιο λογικό τρόπος για την προστασία αυτή είναι να επικεντρώσουμε την αλία στα ποτάμια κυρίως και να την απαγορεύσουμε στην ανοιχτή θάλασσα. Ένα άλλο σχόλιο που δεν άκουσα ακόμη από τους συναδέλφους είναι ότι έχουμε κάποια ποτάμια που στο παρελθόν ε, είχαν ε, πληθυσμούς ε, σολομών, αλλά έχουν βλαβεί από, τα, από υδροηλεκτρικά φαράγματα και έχουν υποβαθμιστεί εκεί οι πληθυσμοί σολομού. Είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα στη Φιλανδία με το πιο σημαντικό ποτάμι Σολομού που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, μπλοκαρίστηκε εξαιτία ενό φράγματο ε, υδροελεκτρικού και έτσι εξαφανίστηκε, εξολοθρεύτηκε εκεί ο, το απόθεμα του Σολομού. Τέτοιου είδου περιπτώσει ε, μπορούμε να τι ανακτήσουμε και να επαναφέρουμε Σολομού σε ποτάμια που στο παρελθόν είχαν τέτοια αποθέματα. Α μην το ξεχνούμε λοιπόν και αυτό. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι τα μέτρα που διευκολύνουν τη διακίνηση ε, των Σολομών είναι σημαντικά, γιατί μερικές φορές φράγματα ή άλλοι λόγοι εμποδίζουν τους Σολομούς να επανέλθουν ε, στα ποτάμια αναπαραγωγής τους. Βέβαια, σε ποτάμια που έχουν εξαφανιστεί τα αποθέματα Σολομού είναι δύσκολο να γίνει ανασύσταση. Αλλά υπάρχουν ποτάμια που εξακολουθούν να έχουν ε, πληθυσμούς άγριου Σολομού. Θα πρέπει να τα προστατεύσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αλία στην ανοιχτή θάλασσα, κατανοώ τα σχόλιά σας, αλλά πραγματικά αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα γενετικά χαρακτηριστικά των αποθεμάτων Σολομών σε συγκεκριμένα ποτάμια, θα πρέπει να περιορίσουμε να απαγορεύσουμε την αλία ανοιχτή θάλασσα. για να επιτρέψουμε την ανασύσταση των αποθεμάτων και πιστεύω ότι αν επιτύχουμε τέτοια ανασύσταση κάποια μέρα θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε και την αλία στην ανοιχτή θάλασσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σάτου Χάση. Ολοκληρώσαμε έτσι τον κατάλογο των ε, ομιλητών και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους εκπροσώπους της Κομισιόν τη Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ. Παρακαλώ. Ε, oui, Καλημέρα σας και ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, εξαιρετική του γραμμαδότηση που πραγματικά ακολουθεί και την ε, δική μας κατεύθυνση. Γιατί ο πρωταρχικός μας στόχος είναι με το πολυευτές αυτό σχέδιο να διαφυλάξουμε τα αποθέματα Σολομού στη Βαλτική και να εξασφαλίσουμε μια ορθολογική και βιώσιμη εκμετάλλευση αυτών των αλληλευτικών αποθεμάτων. Οπότε συμφωνούμε με τη γνωμοδότηση και τη βιβλιοψηφία των τροπολογιών του εισηγητού Βέβαια, υποβάλλοντας την πρότασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη κάποια βασικά πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και κάποια στοιχεία που αναφέρατε κι εσείς στη συζήτηση. Δηλαδή, λάβαμε υπόψη και τον οικονομικό αντίκτυπο των μέτρων που προτείνουμε. Ο εισηγητής βέβαια είναι κάπως πιο φιλόδοξος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το απότερο στόχο. Αλλά εμείς επαναλαμβάνω στις προτάσεις μας λάβαμε υπόψη τα επιστημονικά πορίσματα και τις επιστημονικές γνωματεύσεις. Ό,τι αφορά την ερασιτεχνική ελία και εκεί έχουμε προτείνει κάποια μέτρα για τον έλεγχο και της ερασιτεχνικής αλίας. Ε, μέτρα που ίσχυαν για τον ε, εμπορικό τομέα, για την εμπορική αλλήλεια που αποκομίζει δηλαδή κέρδος οικονομικό από αυτή. Αλλά δεν μπορούμε φυσικά όλα τα μέτρα να τα εφαρμόσουμε και στην αεραστεχνική. Στόχος μας είναι πάντως να εξασφαλίσουμε καλύτερο έλεγχο και της αεραστεχνικής αλλήλειας και συμφωνούμε με τις προτάσεις του εισηγητού. Πάντως εμείς στη δική μας πρόταση λάβαμε ε, υπόψη όλα τα στοιχεία για τη διασφάλιση του αλληλευτικού αποθέματος, για την εξασφάλιση της βιώσιμης εκμεταλλευσής του, με βάση τα επιστημονικά πορίσματα, τις επιστημο... επιστημονικές και προσπαθώντας να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού τις ε, οικονομικές ε, δυσμενείς επιπτώσεις, πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της πρότασής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μοντέση. Ε, και δίνω τέλος το λόγο πάλι στον εισηγητή, τον Καλ Σλίτερ. Ναι, ευχαριστώ την Κομισιόν διότι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Εγώ προχωρώ λίγο πιο πολύ στην ε, πρότασή μου, αλλά πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση και ο στόχος είναι η αποκατάσταση ε, του άγριου σολομού όσο γίνεται περισσότερους ποταμούς γύρω από τη Βαλτική απόλυτα προβλέψιμη είναι ε, η ε, πρόταση η απαγόρευση της ε, αλίας Σολομού στην ανοιχτή θάλασσα είναι όμως και το πιο επίμαχο θέμα. Ε, πρόκειται όμως για οικονομικό πλεονέκτημα, όχι μειονέκτημα. Όλη η Ευρώπη μιλά για ανάπτυξη και μάλιστα βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι ουτοπία, αλλά στις θάλασσες ε, βλέπουμε, ε, βλέπουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Κάθε ε, ψάρι που ε, μεγαλώνει στην θάλασσα μεγαλώνει κατά 15% το χρόνο. Δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση. Το να σταματήσουμε να αλλιεύουμε στην ανοιχτή θάλασσα είναι ε, είναι επένδυση, δεν θα σταματήσει η ε, απλά θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματική. Ε, άλλωστε είναι πολύ πιο οικονομικό και ως προς τον χρόνο και ως προς τα καύσιμα και την ενέργεια ε, και ως προς τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα να λιεύει κανείς κοντά στις θάλασσες αντί να πηγαίνει ε, κοντά στις ακτές αντί να πηγαίνει στην ανοιχτή θάλασσα. Σκοπός είναι δηλαδή να αποκαταστήσουμε τα ε, να αποκαταστήσουμε τα αποθέματα. Θέλουμε να φτάσουμε τους στόχους της ε, Κομισιόν. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τα... Ε, θέλουμε να αποκαταστήσουμε τα αποθέματα. Η πρότασή μου για απογόρευση της αλίας στην ανοιχτή θάλασσα βασίζεται στην επίτευξη της αποκατάστασης των ε, από θεμάτων σολομού στα ποτάμια μας. Ε, αυτό είναι το καλύτερο για όλους, και για τους εραστέχνικους αλείς ε, και τους επαγγελματίες αλληλείς και για την οικονομία. Δεν πιστεύω ότι το 50 και 80% τα νούμερα που αναφέρω εδώ πέρα ότι είναι απλά και ένα λόγια. Εάν ε, αποκατασταθούν τα αποθέματα, ε, δεν θα χρειάζεται να αλλιεύουμε στην ανοιχτή θάλασσα, διότι θα έχουν αποκατασταθεί τα αποθέματα κοντά στις ακτές μας. Ε, και αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικός στόχος και για τους εραστέχνες αλληλείς και για τους επαγγελματίες αλληλείς. Και Χαίρομαι που υπάρχει συμφωνία ως προς τη βελτίωση της υποβολής αναφορών καθώς ε, και για την ε, συλλογή στοιχείων όσον αφορά την ε, ερασιτεχνική αλυσία. Δεν άκουσα παρατήρηση από την Κομισιόν όσον αφορά την, την, την πιο φιλόδοξη πρότασή μου αλλά όπως είπα μπορούμε να σταματήσουμε την αλία στην αριθή θάλασσα αν πετύχουμε αποκατάσταση των αλλιευμάτων. Ε, αν δεν το πετύχουμε αυτό ε, τότε μιλάμε για υποκρισία διότι δύο ποτάμια στην ε, Βαλτική ε, ε, παράγουν το 90% του Σολομού επειδή δεν έχουμε χτίσει εκεί υδροηλεκτρικά εργοστάσια και το υπόλοιπο ε, μεγάλο μέρος του υπολείπου των ε, ψαριών ε, προέρχεται από ένα ποτάμι όπου υπάρχει υδροελεκτρική εγκατάσταση πολύ κοντά στη, στην πηγή του ποταμού και ο υπόλοιπος ποταμός είναι ελεύθερος. Θέλουμε όμως να αποκατασταθεί ο Σολομός σε όσο γίνεται περισσότερους ποταμούς. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε καλό συμβιβασμό όσον αφορά την υποβολή αναφορών. Δεν άκουσα παρατηρήσεις άλλωστε δεν το ανέφερα και ε, ε, νωρίτερα, ε, και για το Σολομό και για την Πέστροφα έχουμε ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης 65 εκατοστό. Ελπίζω όμως... βλέπω ότι υπάρχει βούληση για πρόγραμμα αποκατάστασης και θεωρώ την ε, απαγόρευση που προτείνω για, την απαγόρευση που προτείνω για αλία στην ανοιχτή θάλασσα. Ε, ξέρω ότι είναι ε, επίμαχη, αλλά είναι πολύ φιλόδοξη. Ε, ευχαριστώ τον Καρλ Σλίτερ. Θα ήθελα να ακούσουμε από την Κομισιόν το θέμα σχετικά με το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης. Μιλάμε για περιόδους αποκατάστασης ε, των αποθεμάτων, ε, ε, περιόδους απαγόρευσης αλληλείας και για το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης. Μπορείτε παρακαλώ να απαντήσετε στα θέματα αυτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε. Ε, έχουμε δεχτεί αυτή την τροπολογία για το, ε, το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης. Το σκεφτόμαστε ακριβώς επειδή έχουμε όλο ένα και περισσότερο την εντύπωση πως το ελάχιστο μέγεθος ε, εκφόρτωσης οδηγεί επίσης στην απόρριψη. Είναι ένα θέμα νομίζω που πρέπει να αναλυθεί πιο εις βάθος. Θα μπορούσε να ήταν καλό να θεσπίσουμε ένα μήνυμο, ένα ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης στο σκάφος, ε, γιατί διαφορετικά είναι κάπως πιο περίπλοκο το αναυξήσουμε όμως το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης ε, στη γη, στα λιμάνια, συνήθως οδηγεί σε απόρρεψη. Είναι ένα καλό κριτήριο το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης να χρησιμοποιούμε για την ε, πολιτική μας. Είμαστε ανοιχτοί, θα το αναλύσουμε, αλλά για την ώρα πιστεύουμε πως το μήνυμο μέγεθος εκφόρτωσης οδηγεί στην αύξηση απόρριψης και το ίδιο θα συμβεί και για το απόθεμα Σολομού. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε έτσι την ε, συζήτηση αυτή. Όποιος ε, θέλει να συνεργαστεί ε, για τη γνωμοδότηση αυτή ε, είναι ευπρόσδεκτος. γιατί 27 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και στις 25 Απριλίου θα ψηφίσουμε εδώ την έκθεση του Καρλ Σλούτερ και στην Ολομέλεια προβλέπεται η ψηφορία για τον Ιούλιο του 2012. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε έτσι στο επόμενο θέμα τη ημερησίας διάταξης που είναι το σημείο υπαριθμών 5. Το θέμα εδώ είναι η κοινή αλλιευτική πολιτική. Έχουμε εδώ γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η αρμοδιότητα που μας έχει ανατεθεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, το θέμα είναι λοιπόν πώς φανταζόμαστε το μέλλον της κοινής αλληλευτικής πολιτικής και ε, η συγκητή είναι ο Κρίς Ντέιβις. Παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που μπορώ να σας παρουσιάσω τις προτάσεις μου για την τροποποίηση και τη βελτίωση, ελπίζω, των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή ελευτική πολιτική. Και ως Βρετανός βουλευτής το κάνω αυτό με κάθε ταπεινοφροσύνη, γιατί μόλις την περασμένη εβδομάδα 17 ε, Σκοτσέζοι ε, αλληλεί δικάστηκαν, καταδικάστηκαν ε, γιατί εδώ και κάποια χρόνια ε, αλίευαν το σκουμπρί στην Σκοτία. Δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ήταν φτωχοί, κατακαημένοι που, που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επιβιώσουν. Όμως δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ήταν απλώς λέμαρια, άπλιστοι, πλούσιοι άνθρωποι και πέταξαν ε, στον υπόνομο την καλή φήμη της Βρετανίας. Υπάρχουν ωστόσο αλληλείς που τηρούν τους κανόνες ενώ όλοι οι άλλοι τους καταπατούν. Ε, τους επιβλήθη πρόστιμο 5 εκατομμυρίων ευρώ. Με δεδομένο όμως το τι έκαναν για χρόνια θα έπρεπε να τους έχει επιβληθεί πολύ ψηλότερο πρόστιμο κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής για το μέλλον της, του περιβάλλοντος και της, των μελλοντικών μας αποθεμάτων και θα είναι κρίσιμο το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι αν και η Αλληλευτική Επιτροπή Αλληλείας είναι αρμόδια επί τη ουσία, τα μέλη της Επιτροπής περιβάλλοντο έχουν ρόλο κλειδί να παίξουν για να πείσουν του συναδέλφου ολόκληρο το Κοινοβούλιο να στηρίξουν μεγάλε ε, μεταρρυθμίσεις. Και δεν μπορεί να υπάρχει πιο σαφή ανάγκη. Ο Επίτροπος ε, υπεύθυνο για την Αλληλεία τόνισε ότι το 95% των αλληλευτικών μα αποθεμάτων δεν είναι βιώσιμα στα επόμενα 10 χρόνια, Εκτό και αν γίνουν αλλαγέ. Υπάρχουν δύο θεμελιώδη προβλήματα. Καταρχήν έχουμε μεγάλη υπερβολική και δυνατότητες, πολλά αλλιευτικά σκάφη τα οποία αλλιεύουν λίγα ψάρια και οι Υπουργοί μας έχουν ε, ακολουθήσει μια πολύ κοντόφθαλμη πολιτική. Κάθε χρόνο ε, ε, σαν μονομάχη υποστηρίζουν τα εθνικά τους συμφέροντα και συμφωνούν για όλα ένα και μεγαλύτερα αλλιεύματα. Και τώρα όλοι πληρώνουμε το, το τίμημα ε, στόκ από θέματα τα οποία δεν είναι κερδοφόρα και ένα στόλος ο οποίος μένει ζωντανός μόνο μέσω επιδοτήσεων. Δεν θα πω ότι όλα ήταν τέλεια πριν να έχουμε την ευρωπαϊκή κοινή αλληλευτική πολιτική. Η χώρα μου δεν είναι χαρακτηριστική. Νομίζω ότι ε, φτάσαμε στο αποκορύφωμα των εκφορτώσεων τη δεκαετία του 50 και τότε άρχισαν να πέφτουν κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών όπου μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογράψαμε την κοινή αλληλευτική πολιτική. Ε, κάναμε καλή δουλειά καταστρέφοντας τα δικά μας τα ηλεκτρικά αποθέματα οι ίδιοι. Η ΚΑΠ δεν βοήθησε για πολλά χρόνια, αλλά για να είμαστε δίκαιοι η κατάσταση είναι πιο σταθερή αυτή τη στιγμή και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν και κάποιες επιτυχίες. Όπως για παράδειγμα στον Ατλαντικό μια μεγάλη ανάκαμψη των στόκ ε, ε Έχουμε δει επίση ε, το ίδιο στη Βαλτική και αυτό έχει επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της Βαλτικής ε, έχουν γίνει καλά πράγματα και η Κομισιόν προτείνει πολύ σημαντικές αλλαγές. Θέλει να θεσπίσει πλάνα σχέδια διαχείρισης για κάθε αλίευμα. Το στόχος είναι να επιτύχουμε πάνω από την βιώσιμη το ε, απόθεμα μέχρι το 2050. Είναι αυτό εφικτό. Σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μέχρι 80% των ε, ψαριών που λαλιεύουν ή αλληλείς ε, πετιούνται στη θάλασσα νεκρά. Αυτό δεν είναι απλώς κακές, κακή επιχείρηση. Θα έπρεπε να είναι και ανήθικο. Η Κομισιόν θέλει να πετύχει μειώσεις στις ε, δυνατότητες και να προωθήσει και νέες επιχειρήσεις ε, έτσι ώστε να υπάρχουν ε, δυνατότητες μεταφοράς των επιχειρήσεων. Παρόμοια προγράμματα έχουν γίνει στη Δανία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστρία, στην, στην ΣΥΠΑ και θα ήθελε τα περιφερειακά όργανα να κάνουν τη διαχείριση και όχι Βρυξέλλες. Ορισμένοι διαμεμαρτύρονται ότι οι προτάσεις στον κανονισμό δεν είναι αρκετά συγκεκριμένες, αλλά είναι μια διαδικασία από κάτω προ τα πάνω. Τα περιφερειακά σώματα θα πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να πούν τι επιθέμουν. Η Κομισιόν θέλει επίση να προωθήσει τι υδατοκαλλιέργειε και στι χωριστέ προτάσει ζητά πολύ πιο υψηλέ προδιαγραφέ για τα αλλιευτικά σκάφη τη Ευρώπη που αλλιεύουν σε αλλοδαπά ύδατα και Επίση, θέλει να σταματήσει τι επιδοτήσει για διάλυση σκαφών, όπου όπω είδαμε στην πρόσφατη έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου έχουν κοστίσει τεράστια ποσά, αλλά δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν τι δυνατότητε των αλευτικών μα στο Αντί γι' αυτό θα έπρεπε τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν ώστε να βοηθήσουν του αλληλεί να ανταποκριθούν στις απαιτήσει και να βοηθήσουν τι παράκτιες κοινότητε να προσαρμοστούν σε αλλαγέ. Εγώ πιστεύω πω η πρόταση είναι ριζική και ισχυρή και θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική στην αποκατάσταση των αποθεμάτων και αξίζει να τη στηρίξουμε. Εγώ έχω καταθέσει πάνω από 100 τροπολογίες, αλλά ο είναι να συμπληρώσουν και να βελτιώσουν τις προτάσεις τη Κομισιόν, καθώς και να γεμίσουν κάποια κενά και νομίζω ότι εν γέννη θα υποστηριχθούν και από την Κομισιόν. Ε, εν συντομία, αυτό που θέλω να κάνω είναι να τεθεί στην καρδιά της πολιτικής μας ε, ε, την υγεία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τα υγιή ψάρια είναι το καλύτερο για μας. Θέλω να ξεπεράσουμε τα μήνυμα κριτήρια για την βιώσιμη αλία. Αυτό θα σήμαινε <clears throat> να σταματήσουμε την αλία, να μειώσουμε τη θνησιμότητα των ψαριών. Να μπορούν δηλαδή τα ψάρια και η αλευτική μας βιομηχανία να είναι υγιής. Δεν θέλω μόνο πολλά ψάρια, θέλω πολλά μεγάλα ψάρια. Στην χτεσινή ε, συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Αλληλείας, ο Επίτροπος Αλληλείας είπε στους εθνικούς βουλευτές ότι στη Μεσόγειο αυξάνεται η αγορά για μικρά ψάρια και οι αλληλείς επίτηδες αλλιεύουν ψάρια που είναι πολύ νεαρά για να αναπαραχθούν. Μα αυτό είναι τρελό. Πριν, <laughs> πριν να τα ψαρέψουμε, ας αφήσουμε τα ψάρια να έχουν σεξουαλικές επαφές. Ένα τέτοιο σλόγγαν θα πρέπει να υιοθετήσουμε ε, για όλα τα ψάρια, όλα τα είδη, όχι μόνο τα εμπορικά. Να, τους αφήσουμε, να τα αφήσουμε λοιπόν να επιβιώσουν. Νομίζω πως υπάρχει μεγάλη συνένεση στο Κοινοβούλιο και σίγουρα στην, Αλία, στην Επιτροπή Αλίας ότι οι απορρίψεις θα πρέπει να απαγορευτούν ανά είδος, ανά αλίευμα με προτάσεις που θα μπουν μέσα στα προγράμματα τα μακροπρόθεσμη διαχείριση. Οι αλληλείς λένε ότι ναι θέλουν να σταματήσουν απορύψα, αλλά δεν είναι πρακτικό κάτι τέτοιο. Μόνο άμα κάνουμε όμως, εισάγουμε απαγόρευση θα πετύχουμε κάτι. Ε, γιατί έτσι θα σταματήσουμε και με τις, αυτές τις ιστορίες με το πιο, επιλεκτικά, πιο επιλεκτικό εξοπλισμό κτλ. Θα υπάρξει ανάπτυξη ενός εξοπλισμού που θα ανταποκρίνεται στην απαγόρευση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να φτιάξουν τέτοιες πολιτικές, ε, πρέπει να το έχουν κάνει εδώ και χρόνια και αυτό πρέπει να αλλάξει. Εγώ προτείνω και για τα κράτη-μέλη που δεν κάνουν τη δουλειά τους καλά. Ε, επειδή οι ευρωβουλευτέ είμαστε συνομοθέτε εδώ, θα πρέπει να έχουμε τελικό λόγο για κάθε μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διαχείρισης, αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει κάποιες ποσοστώσεις για το Συμβούλιο περισσότερες. Πώ λοιπόν θα περιορίσουμε του υπουργού και πώ θα του αναγκάσουμε να λάβουν υπόψη τι συμβουλέ μα. Η νομική υπηρεσία μας, ε, μου έδωσε κάποιε συμβουλέ και ελπίζω πω κάποιε υπερβολογίες μου θα λύσουν αυτό το ζήτημα. Τώρα υπάρχει μεγάλη αντίρρηση όσον αφορά τι άδειε αλίευση και τη δυνατότητα μεταφορά αυτών. Εγώ νομίζω πω είναι λάθο αυτό. Δεν θα υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα υπάρξουν 27 διαφορετικά. Καθένα από αυτά θα τα έχει συντάξει ο εκάστοτε κράτο μέλο. και θα λαμβάνει υπόψη τις εθνικές ε, ανησυχίε και προβληματισμούς. Αν θέλουν να βοηθήσουν του αλληλείς μικρή κλίμακα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι μόνο οι ενεργοί αλληλείς θα ε, έχουν τι άδειε και όχι οι ποδοσφαιρικές ομάδες ε, και οι λέσχε διαφόρων ηθών και αν φοβούνται μήπως πολύ λίγοι μαζέψουν στα χέρια τους όλη την αλία, τότε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να το αποφύγει, αν μια κυβέρνηση αυτό επιθυμεί. Και λέω στις τροπολογίε μα τρόπους για να ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι κυβερνήσει για να περιορίσουν τα πράγματα. Αλλά είναι πολύ εύκολο οι κυβερνήσει να τα ρίχνουν όλα στι Βρυξέλλε και να μην αναλαμβάνουν τι ευθύνε του, αλλά εγώ δεν νομίζω θα πρέπει να του διευκολύνουμε. Η κάλπη μπορεί να αποτελέσει τη λύση για πολλά από τα προβλήματα και παρά τα όσα λένε κάποιες ε, ΜΚΟ, αλλά όχι όλε, δεν υπάρχουν πολλέ εναλλακτικέ που να λειτουργούν. Και το πρόβλημα είναι κατά τη γνώμη μου, ε, οι άνθρωποι αυτοί που είναι έτοιμοι να διχάσουν την μάλλον να, να φτιάξουν μια τέτοια κάπ, κάλπ που να ανταποκρίνεται σε όλα αυτά. Ε, ένα πρόβλημα από αυτά είναι η μικρή κλίμακα αλληλεία. Το 70% των θέσεων απασχόληση είναι αυτή η μικρή κλίμακα αλληλεία. Και ο αντίκτυπο στην αλληλεία, στο περιβάλλον, με συγχωρείτε, είναι μηδαμινό. Τα κράτη-μέλη, ωστόσο, θα πρέπει να ε, χορηγήσουν τις ποσοστώσεις. Η χώρα μου ε, δεν τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Ενώ δίναμε ας πούμε 40% των ποσοστώσεων στους μικρούς ε, αλληλείς. Ε, στην Σουηδία για παράδειγμα η ποσόστοση αυτή ήταν 20%. Και εν τέλει τα πάντα για την αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να είναι διαφανή και ανοιχτά γιατί ε, στο κοινό. Να μην κρύβει κανείς δηλαδή τι ψαρεύει. Και έχω υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Ολόκληρο το κοινοβούλιο όλοι λένε πως θέλουν βιώσιμη αλληλευτική πολιτική. Στην πράξη όμως η Κομισιόν έχει να αντιμετωπίσει πολύ στεναρή αντίρρηση από πολλά κράτη-μέλη που θέλουν να μπλοκάρουν τη μεταρρύθμιση και να συνεχίσουν όπως μέχρι τώρα ε, και κυβερνήσεις ε, που αντιστέκονται. Όμως θα πρέπει να ιτηθούν αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμα αλλιευτικά αποθέματα. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει εμείς εδώ σε αυτή την Επιτροπή να πιέσουμε για ριζικές αλλαγές στην αλλιευτική πολιτική. Είναι πολύ εύκολο να επικρίνουμε, αλλά τώρα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις και όσοι δεν, σε όσους δεν, αρέσει, δεν αρέσουν οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλουν συγκεκριμένες τροπολογίες, εναλλακτικές λύσεις. Και θα πρέπει να δούμε και εκείνους Επιτροπή κανονικά και φυσιολογικά δεν ενδιαφέρονται για την αλληλεία και βλέπω εδώ τον ε, κύριο Σέιμορ ε, που είναι από την Αυστρία που δεν είναι γνωστή για τον αλληλευτικό της στόλο αλλά θέλουμε τη στήριξη ακόμα και των κρατών που δεν έχουν αλληλευτικούς στόλους για να έχουμε όλοι ψάρια και να φάμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν υπάρχουν ψάρια δεν θα υπάρχουν και ε, ψαράδες και δεν χρειάζεται να είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να πάψουμε να υπονοούμε τις αποδείξεις που υπάρχουν, τις ενδείξει που υπάρχουν, να φτιάξουμε πολιτικές που είναι σωστές για το μακροπρόθεσμα. Αν το κάνουμε αυτό μπορούμε να έχουμε υγιεί θάλασσε, επιτυχή βιομηχανία και ένα σωρό ψάρια, μπόλικα ψάρια για το μέλλον. Ευχαριστώ, πολύ. Κρίς Ντέιβις, έχει έρθει η ώρα της απόφασης. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε πώς, τι θα αποφασίσουμε. Έχει καταρχήν το λόγο ο Κρίστοφερ Φιέλνερ, παρακαλώ, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Κρίς. Η εντύπωσή μου για τον Κρίς είναι σε μεγάλο βαθμό ότι είναι πολύ μελοδραματικός, ε, είναι ακραίος ε, και υπερβάλλει. Αυτή τη φορά όμως έχει δίκιο και μάλιστα πολύ δίκιο. Ε, έχω συμμετάσχει σε πολλές ε, συζητήσεις ε, όπου σκέφτομαι, σκέφτομαι όχι πάλι τα ίδια λέει, αλλά αυτή τη φορά έχει δίκιο και χαίρομαι που έχει αναλάβει αυτό το θέμα για την Επιτροπή μας. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα είπες, διότι συμφωνώ με σχεδόν όλα. έχω την εντύπωση όμως ότι αν δεν κάνουμε τη δουλειά σωστά αυτή τη φορά δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Η Επίτροπος Αλίας, η κυρία Ταμανάκη, όταν μας λέει ότι το 91% των αποθεμάτων ε, μπορεί να εξαντληθούν σε 10 χρόνια ε, εάν ε, δεν κάνουμε κάτι σωστό αυτή τη φορά. Έχει δίκιο και... Ανέφερε στο παράδειγμα του γάδου στη Βαλτική θάλασσα. Πριν κάποια χρόνια στη Σουηδία είχαμε συζήτηση για το αν θα πρέπει να απογορευτεί η αλία του γάδου στη Βαλτική θάλασσα, διότι πιστέψαμε ότι μπορεί να εξαφανιστεί τώρα θεωρείται ότι είναι βιώσιμο το απόθεμα αυτό και αυτό είναι το αποτέλεσμα πολιτικών, ε, ενός σχεδίου διαχείρισης, των σωστών πολιτικών. Και ε, γι' αυτό ακόμα και σε αυτή τη δραματική κατάσταση ε, ε είμαι αισιόδοξο, διότι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Νομίζω το, το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει η Επιτροπή μα είναι να υποστηρίξει την πρωτοβουλία της ε, Επιτρόπου και της Κομισιόν, διότι με την ευρεία έννοια κινεί την πολιτική προ τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι οι προσθήκε σου γενικά ε, αξίζει να υποστηριχθούν. Εγώ θα ε, ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Καταρχήν την περιφερειοποίηση, διότι πιστεύω ότι παρότι ε, μιλάμε για τεχνικό επίπεδο και νομικές πτυχές, είναι σημαντικό να αυξήσουμε την νομιμότητα της πολιτικής. Οι συμμετέχοντες να ε, έχουν την αίσθηση ότι οι κανόνες διαμορφώνονται με τρόπο που να προσαρμόζονται στην πραγματικότητά τους, διότι αν δεν το πετύχουμε αυτό, ε, ο κόσμος δεν θα συμμορφωθεί με τους κανόνες. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η περιφερειοποίηση. Δεύτερον, όσον αφορά τις μεταβάσιμες ε, ποσοστώσεις αλληλείας. Πιστεύω ότι είναι καλό ότι πιστεύεις ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το εφαρμόσουν. Το πώς θα εφαρμοστούν αυτά ε, όμως θα πρέπει να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Είχαμε αρκετά προβλήματα παροπλισμού για τα σκάφη αλίας ε, και τελικά τα βλέπουμε να εμφανίζονται αλλού και ε, λαμβάνουν νέε επιδοτήσεις σε έναν τομέα που ούτως ή άλλως λαμβάνει υπερβολικές επιδοτήσεις αλλά οι μεταβάσιμες ε, αλλιευτικές ε, παραχωρήσεις ε, φαίνεται να είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο. Και σχεδόν όλα τα προβλήματα που έχουμε από περιβαλλοντικής πλευράς είναι ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για κάτι που δεν τους ανήκει. Είτε μιλάμε για νερό, είτε για αέρα, είτε για αποθέματα αλληλείας. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για κάτι που δεν τους ανήκει. Εάν όμως μιλάμε για παραχωρήσεις και, ε, τις, ε, και τους ανήκουν αυτές, ε, τότε θα ενδιαφερθούν. Και, νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τις αλληλευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. έχουν βελτιωθεί τον τελευταίο καιρό. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι η βασική μας ιδέα θα πρέπει να είναι ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει, ψαράδες θα πρέπει να τηρούν τους ίδιους κανόνες οπουδήποτε και να λιεύουν. Ιδιαίτερα εφόσον εμείς οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι πληρώνουμε γι' αυτό και αναγοράζουν ε, ψάρια αλλού θα πρέπει να αναλάβουν τις ίδιες περιβαλλοντικές ευθύνες και αλλού. Σαν να βρίσκονταν εδώ, εντός της Ευρώπης. Δεν έχω τόσες πολλές τροπολογίες, να σκέφτομαι αλλά κυρίως στον τομέα της εγγύησης και της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ώστε να πούμε δηλαδή πως τα κράτη-μέλη εκεί που ε, υπάρχει κοινή αλληλευτική προσπάθεια να συνεργάζονται σε αυτήν. Εκεί σκοπεύω να κάνω κάποιες τροπολογίες. Πιστεύω πως το πιο σημαντικό όμως είναι να φροντίσουμε ώστε αυτή η Επιτροπή όχι επισήμω να αναλάβει την ε, έκθεση επί της ουσίας, αλλά ηθικώς ναι. Γιατί πολύ μικρή είναι η ομάδα των πολιτικών στα κράτη-μέλη και σε αυτό το κοινοβούλιο που έχουν ασχοληθεί με την αληφτική πολιτική και ε, ήταν πολύ αρνητικό αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερους υπουργούς, υπουργούς αλληλεία στα κράτη-μέλη και περισσότερους ευρωβουλευτές και όχι μόνο αυτούς τη αλληλείας για να ελέγχουμε τις, ε, την, τις ε, αντιδράσεις τους. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό θα συνεχίσουν ε, τα ίδια παντελάκι μου και δεν πρόκειται να α, πετύχουμε τίποτα. Ευχαριστούμε κύριε Φιέλλερ. Η κυρία Λίντα Μακέβεν και μετά Eckhout. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον Κριστοφέρο ότι είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτό το δεύτερο μισό της Κοινοβουλευτικής θετίας της Επιτροπής μας. Δεν ήθιστε μια γνωμοδότηση να έχει τέτοια σημασία, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε συναπόφαση για τα θέματα αυτά και συμφωνώ απόλυτα ότι χρειαζόμαστε ευρεία συζήτηση για το θέμα αυτό. Παρά ήταν βολικό και για τους υπουργού και για τους αλληλείς και για τις ελευτικές κοινότητες να κατηγορούν την ΚΑΠ, την ελευτική πολιτική και τις Βρυξέλλες για τα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι με την νέα νομοθεσία όλοι θα έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν ε, τις ευθύνες τους, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να συναποφασίσουν στην ε, κατάλληλη κοινή ελευτική πολιτική για την Ευρώπη. Και οι κυβερνήσεις και οι ελευτικές κοινότητες θα έχουν το λόγο τους στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής. Συμφωνώ με την πλειονότητα των τροπολογιών του ΚΡΙΣ και συμφωνώ επίσης ότι το πιο σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε τα λευτικά αποθέματα για το μέλλον και η διαχείρισή τους να στηρίζεται σε ανεξάρτητα επιστημονικά απορίσματα και όχι μόνο σε αιτήσια παζαρέματα στο Συμβούλιο Υπουργών Συμφωνώ λοιπόν με τις τροπολογίες που έχουν αυτό το χαρακτήρα, αυτή την κατεύθυνση. Να είμαστε αυστηροί για τις απορρίψεις. Μου λένε ότι είναι περίπλοκο το θέμα. Πάντως είναι ρεαλιστική η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πού είναι η εναλλακτική λύση. Όσοι λένε ότι δεν θα λειτουργήσουν οι απαγορεύσεις των απορρίψεων, ας μου πούν ποια είναι η εναλλακτική λύση. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι αποτελεσματική αυτή η πρόταση. Άλλωστε εναλλακτική δεν υπάρχει. Πολύ συχνά στη δική μου πατρίδα είχαμε μία εκστρατεία από ένα γνωστό σεφ που έλεγε ε, απαγορεύσε τις απορρίψεις. Τώρα αυτοί που έλεγαν πέρυσι απαγορεύσεις φέτος διαφωνούν. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση, πώς θα διαφυλάξουμε διαφορετικά τα ελευτικά μας αποθέματα. Σε ό,τι αφορά τις μεταβιβάσιμες αλληλευτικές άδειες. Και αυτό το θέμα προκαλεί σφοδρή συζήτηση και θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή. Πάντως το μέχρι τώρα σύστημα τουλάχιστον πατρίδα μου είναι αδιαφανές. Δεν μπορεί η κυβέρνηση σήμερα να πει ποιος είναι ο δικαιούχος της ελληνικής άδεια. Δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των, της άδειας. 96% των αδειών κατέχονται από 23 ενώσεις παραγωγών και μόνο 4 με 6% ανήκουν σε μικρούς σε μικρών αλληλευτικών κοινοτήτων ε, για τις οποίες ακούμε πολλά και διαρριγνούμε τα μάτια μας για αυτές. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν τις άδειες. Και όσοι θέλουν περισσότερε άδειε πρέπει να πληρώσουν στι ε, οργανώσει αλλαίων. Θα δούμε λοιπόν να αναθεωρήσουμε το σύστημα των μεταβιβάσεων αδειών. Ακούσαμε ότι ακόμη και ποδοσφαιρικοί σύλλογοι έχουν τέτοιε άδειε αλλιευτικέ. Λένε ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί αυτό για του ποδοσφαιρικού ομίλου. Αλλά να δούμε. Ποιοι έχουν πραγματικά, ποιοι είναι οι κύριοι αυτών των ε, αδειών. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια για το σύστημα και είναι που δεν γνωρίζουμε ποιο κατέχει αυτά τα αλληλευτικά δικαιώματα. Οπότε ένα σύστημα μεταβιβάσεων αλληλευτικών αδειών θα πρέπει να στηρίζει σε πολύ διαφορετική βάση από τη σημερινή. Επίσης ε, θέλουμε ένα σύστημα που θα επιβραβεύουμε τους ε, έντιμους και σωστούς ελείς. Αναφέρθηκε ε, η εγκληματική δραστηριότητα πολλών εκατομμύριων στερλινών. 16 εκατομμύρια όμως. είπατε 59. Ε, πού οφείλεται αυτή η διαφορά. Πάντως όντως υπάρχει και παράνομη αλεία. Αλλά μερικοί είναι και έντιμοι. Θα πρέπει το σύστημα να επιβραβεύει τους έντιμους αλείς, τους σωστούς. Θέλουμε βιωσιμότητα, θέλουμε να βοηθήσουμε τους αλείς που θα συμβάλλουν σε αυτή την εξασφάλιση της αηφόρου αλείας. Επίσης το θέμα της περιφερειοποίησης, αποκέντρωσης του συστήματος. Συμφωνώ με την ιδέα της αποκέντρωσης. Αλλά δεν φαίνεται από την νομοθεσία πώς θα λειτουργήσει το σύστημα με σαφήνεια. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν είναι ρητή νομοθεσία θα μπορεί εύκολα κανείς να την παρακάμψει. Αναφέρεται η ανάγκη αιτήσεων πολιετών μάλλον σχεδίων. Αλλά πώς θα ισχύσουν αυτά τα πολιετή σχεδιαδράσεις. Φαντάζομαι ότι είναι διαπεριφερειακά, ένα για τη Βαλτική, ένα για τη Βόρεια Θάλασσα, αλλά ποιος θα είναι ο προτεργάτης ενός τέτοιου σχεδίου. Ποιο θα χρηματοδοτήσει τι γραμματείε που θα συντάξουν τα σχέδια, ποιε είναι οι προθεσμίε για την υποβολή των σχεδίων, πώ θα γίνεται η αστυνόμευση και ο ελεγχό του, πώ θα λειτουργήσουν σε, στα πλαίσια μια συνθήκη που μπορεί να ελέγξει μόνο τα κράτη-μέλη, το κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει αυτό να το προσδιορίζουμε σε τροπολογίε, θα πρέπει πιο λεπτομεριακά να προβλέπετε στην νομοθεσία. Φοβάμαι μη θα σπίσουμε μια νομοθεσία και μετά από δύο χρόνια να μα πει κάποιο. ναι αλλά ποιο έχει την πρωτοβουλία για τα σχέδια, ποιο θα τα υποβάλει, θα τα επιβλέπει η κεντρική διοίκηση των Βρυξελών. Όλα αυτά θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στην νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε τι παράκτητες κοινότητε με κάποιο τρόπο. Και πολλοί μιλάνε για την αλληλευτική βιομηχανία στις παράκτιες κοινότητες. Νομίζω όμως ότι τα περισσότερα, οι περισσότερες βιομηχανίες δεν επενδύουν στις παράκτιες κοινότητες. Τα περισσότερα εργοστάσια μεταποίησης βρίσκονται μακριά από τις παράκτε κοινότητες. Συμφωνώ λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε τις επενδύσεις στις παράκτιες κοινότητες. Κάτι που μέχρι τώρα δεν αναφέρθηκε και ίσως δεν έχει το θέση σε αυτή την νομοθεσία Πάντως μας ενδιαφέρει. Οι εργασιακές συνθήκες αυτών που απασχολούνται στην αλία, στον κλάδο αυτό. Γιατί μιλάμε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε τις θέσεις απασχόλησης, αλλά ποιο ποσοστό όσων εργάζονται στα ληφτικά σκάφη προέρχονται από τρίτες χώρες. Από την Ινδία, από τις Φιλιππίνες, άνθρωποι που επειδή εργάζονται στην ανοιχτή θάλασσα στα σκάφη, δεν λαμβάνουν τον ελάχιστο βρετανικό μισθό, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία. Λαμβάνουν μισθούς πείνα και έρχονται για λίγους μήνες, εποχιακά επιστρέφουν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα υγεία ή δεξιδοτικό. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως να ρυθμίσει την κατάσταση, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει. Και το αγνοούμε αυτό πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πολύ συχνά έχουμε εργαζόμενους αλλοδαπούς ε, που δεν ε, τους επιτρέπεται καν να αποβιβαστούν για να εξασφαλιστούν αυτές οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες μόνο και μόνο επειδή εργάζονται στα σκάφη και στην ανοιχτή θάλασσα. Τίποτα δεν γίνεται για να βοηθήσουμε βελτίωση κατάσταση, αλλά έτσι δεν ε, εξυπηρετούμε και την απασχόληση στις δικές μας κοινότητες. Θα είναι πραγματικά η λίθος ε, αυτή η νομοθετική προσπάθεια, γιατί για πρώτη φορά έχουμε συναπόφαση σε αλληλευτικά θέματα. Δεν υπάρχουν λοιπόν, δεν έχουμε άλλα προσχήματα, μορφές και κατηγορίες προς την Επιτροπή από τους ε, υπουργού για, ε, για το παζάρεμα που γίνεται κάθε χρόνο για την καταχώρηση των κατανομή των ποσοστώσεων. Δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες και προσχήματα θέλουμε διαπραγμάτευση με όλους, γιατί σε τελική ανάλυση, αν δεν εξασφαλίσουμε βιώσιμο κλάδο αλίας, και ακούω ήδη τις αντιρρήσεις, θα μας πει το Συμβούλιο ότι δεν αρκεί κανείς ε, να πούμε στο Συμβούλιο δεν αρκεί κανεί να διαφωνεί με την Επίτροπο Δαμανάκη. Εναλλακτικέ λύσει έχετε, εναλλακτικέ προτάσει έχετε, ποιε να τι εξετάζουμε. Δεν αρκεί να μα λέτε δεν μα αρέσουν ε, οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταθέστε μια εναλλακτική πρόταση, μπορεί να είναι καλύτερη. Αλλά όχι μόνο αρνητικότητα και διαφωνία. Γιατί μερικοί θεωρούν ότι μια παρελκυστική τακτική, μια καθυστέρηση της πρώτης ανάγνωσης στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ε, θα κερδίσουν χρόνο και θα τορπιλήσουν το σύστημα. Να μην επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε για την αναθεώρηση της κοινή ελευτικής πολιτικής από την ε, εποχή που πρωτοίσχυσε. Νομίζω ότι θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Λίντα Μακέβαν. Για τους πράσινους... Οι πράσινοι τώρα παίρνουν το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Κρίση, για την έκθεσή σου για το σημαντικό αυτό θέμα. Ας ελπίσουμε πράγματι ότι θα αναλάβουμε την ευθύνη Λίντα, διότι συμφωνώ ότι αυτή είναι η ευκαιρία και η στιγμή να ε, ε, ε, ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όμως να μην το αφήσουμε το θέμα αυτό αποκλειστικά στην ε, Επιτροπή ε, Αλίας, όπως δεν πρέπει να αφήσουμε και τη συζήτηση περί Γεωργίας αποκλειστικά στην Επιτροπή Γεωργίας, ε, διότι τότε δεν νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να επιφέρουμε τις αλλαγές που είναι απαραίτητες και στις δύο μεταρρυθμίσεις. Κρίση, σε ευχαριστώ πολύ για την εκθεσή σου. Η πράσινη μπορούν να την στηρίξουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά αυτό που είπες για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και την προστασία των ε, θαλασσίων οικοσυστήματων είναι πολύ σημαντικά. Δύο σημαντικά θέματα όμως απομένουν να συζητηθούν και θα πρέπει να ε, τα εξετάσει η Επιτροπή μας. Ε, η ικανότητα του στόλου και οι μεταβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις. Νομίζω ότι αυτά τα δύο θέματα θα γίνουν πολύ σημαντικά. Καταρχήν η ικανότητα του στόλου. Αυτό δεν αναφέρθηκε αρκετά μέχρι τώρα, αλλά αυτό είναι το, το πρόβλημα. Έχουμε πολλά, πολύ μεγάλα σκάφη, ε, υπερβολικά πολλά, υπερβολικά μεγάλα σκάφη, τα οποία ε, αλλιεύουν. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και σκέφτομαι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι στην έκθεσή μας, διότι είναι πράγματι ε, ζωτικής ε, σημασίας και θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις σχετικά με το πόσο, πόσα σκάφη υπάρχουν, ποιες είναι οι επιπτώσεις τους ε, στην υπεραλίευση, ποια, ποια σκάφη είναι ε, τα πιο καταστροφικά. Θα πρέπει να ε, προωθήσουμε τα σκάφη τα οποία είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Θα χρειαζόμαστε λοιπόν όχι μόνο ανάλυση αλλά και προγράμματα μείωσης του στόλου και θα πρέπει να δούμε ποια σκάφη πρέπει να παροπλιστούν πρώτα. Επίσης ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, προσέξουμε περισσότερο την ε, ικανότητα του στόλου στα πολυετή προγράμματα θα πρέπει να ε, ε, εξεταστεί η ικανότητα του στόλου σε σχέση με τα αλλιευτικά αποθέματα και θα πρέπει ε, να υπάρξουν προγράμματα για τη μείωση του, της ικανότητα ικανότητας που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει στα πολιετή πλαίσια, αυτό, πολιετή προγράμματα. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό θέμα και θα ασχολούμαι με αυτό, η ικανότητα του στόλου δηλαδή. Δεύτερον, με μεταβάσιμες αλλιευτικές παραχωρήσεις. Είναι, γίνεται πολύ έντονη συζήτηση, το γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα ε, είναι μια συζήτηση που έχει τα στήματα και ε, γνωρίζω και τον Κρίσε και τον... Ε, και, κύριε Φιέλνερ, μπορεί, μπορεί ε, μερικές φορές να υπερβάλλει, αλλά έχει δίκιο και πάντα είναι πολύ με, μετριοπαθής στην συζήτηση στο τέλος. Ε, ξέρω ότι γνωρίζετε ε, τις θέσεις πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων, ταυτόχρονα όμως να ε, ισχυρίζεται κανείς ότι οι με αλληλευτικές παραχωρήσεις μειώνουν την, τον, την αλληλευτική ικανότητα, αυτό είναι ανοησίες, το γνωρίζετε, δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα, ένα από αυτά είναι η, η μεγάλη ικανότητα του στόλου και Και ξέρουμε ότι οι μεταβάσιμε αλληλευτικέ παραχωρήσει δεν μειώνουν την αλληλευτική ικανότητα. Ε, παράδειγμα, οι κάτω χώρε όπου έχουμε αυτέ τι μεταβάσιμε ποσοστώσει και έχουμε ακόμα το πρόβλημα τη υπερβολική αλληλευτική ικανότητα. Ε, και στο στι κατοχώρε. Ε, εάν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, μην ισχυρίζετε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τι μεταβάσει μα ελευθερικέ παραχωρήσει. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει και μια πολύ βασική ε, συζήτηση σχετικά με το πώ βλέπουμε τα ψάρια. Πρόκειται για ε, εμπόρευμα ή πρόκειται για φυσικό πόρο. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για δημόσιο φυσικό πόρο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ε, όταν ε, εμποροποιούμε αυτό τον πόρο με, τα, ε, με τις μεταβάσιμες ποσοστώσεις. Εάν επίσης κάνουμε υποχρεωτικές τις μεταβάσιμες ποσοστώσεις, αυτό θα είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε πολύ περισσότερο στο δικαίωμα αλληλείας και μάλιστα με βιώσιμο τρόπο. Ε, αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης και κατόπιν θα μπορούμε να ε, κοιτάξουμε τα κριτήρια. Η αλία να συμβάλλει στην τοπική οικονομία. Ε, τα εργαλεία να είναι σωστά, να μειωθούν οι απορρίψεις, να εξετάσουμε τη, τη ζημιά του βυθού ή κατανάλωση καυσίμων, αλλά και το αν πρόκειται για νόμιμη ή παράνομη αλληλεία θα Πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα κριτήρια ώστε ο κόσμος να έχει το δικαίωμα να αλλιεύει ε, με τρόπο ε, κοινωνικά και ε, περιβαλλοντικά βιώσιμα. Πάντως εγώ δεν έχω πιστεί ότι οι μεταβάσιμες αλληλευτικές ποσοστώσεις θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά χαρακτήρα, διότι μέχρι τώρα έχουμε δει πολλά προβλήματα σχετικά με τον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί αυτές οι μεταβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις. Και αν δεν ασχοληθούμε πρώτα με τα προβλήματα αυτά, δεν θα πρέπει να ε, κάνουμε υποχρεωτικό το στοιχείο αυτό στα πλαίσια ενό νέου συστήματο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο επικριτικοί, πολύ πιο προσεκτικοί και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια ει συζήτηση για το θέμα αυτό. Εάν όμω ε, τελικά εμεί από την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ασχοληθούμε με την ικανότητα του στόλου από τη μία και ε, από την άλλη ε, επιδιώξουμε μια πολύ καλύτερη συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων, τότε νομίζω ότι θα δώσουμε κάτι που θα βελτιώσει τις αλληλευτικές πολιτικές. Προσβλέπω σε μια πολύ καλή επικοδομητική συζήτηση με τον Κρι και του άλλου ε, και ε, στην υποβολή προτάσεων που πραγματικά θα επιφέρουν σημαντικέ αλλαγέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Άικχαουτ. Ε, ο Μάρτιν Κέλεμαν για, για την πολιτική ομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη ε, από τη Σκιώδη Σίτρια που δεν μπορεί να είναι παρούσα και μου ζήτησε να πω λίγα λόγια εκ μέρους της. Ε, να ευχαριστήσω τον Κρίς για την δουλειά που έχει κάνει στο θέμα αυτό. δεν θα συμφωνήσω με τον προλήσαντο ότι έχει δίκιο σε όλα, αλλά σίγουρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο ε, καθήκον να συμβάλλουμε ε, στο να διαμορφωθεί σωστά η αλληλευτική πολιτική. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα εδώ τα οποία ε, θα πρέπει να ξεπεράσουμε, να καταπολεμήσουμε, ιδιαίτερα στην Επιτροπή Αλίας. Στόχος μας είναι λοιπόν να οδηγήσουμε την πολιτική αυτή προς τη σωστή κατεύθυνση. Να ξεκινήσω με την αναγνώριση ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική μέχρι τώρα, όπως είπαν και άλλοι, προσπάθησε να μετριάσει την ε, περιβαλλοντική καταστροφή. Έχει αποτύχει όμως. Ε, έχει ε, αποτύχει η μικροδιαχείριση. Η υπεραλίευση είναι πολύ ευρύ φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποθέματα μας έχουν γίνει ιδιαίτερα ευάλωτα. Γι' αυτό η ομάδα μας, όπως και οι περισσότεροι από άλλους που πήραν το λόγο σήμερα, θέλουν μια πραγματική μεταρρύθμιση ώστε να πετύχουμε υγιή αποθέματα και μια καλή αλλιευτική βιομηχανία και ένα ε, καλό θαλάσσιο περιβάλλον. Η μεταρρύθμιση της κοινής αλλιευτικής πολιτικής μας δίνει ε, μια ε, ευκαιρία που μας δίνεται μια φορά ανά να αντιμετωπίσουμε το θέμα των απορρίψεων, εξαλείψουμε την ε, μη αποτελεσματική μικροδιαχείριση ε, και να ε, καταργήσουμε και τους κανόνες περί ποσοστώσεων που δεν λειτουργούν καλά. Η Κομισιόν προτείνει διάφορα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν και πολλά περισσότερα που μπορούμε να προτείνουμε για να πετύχουμε μια καλύτερη πολιτική. Για την υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να ασχοληθούμε με την εξάρτησή μας από, από τα εισαγόμενα τρόφιμα. Θα πρέπει να στηρίξουμε ακολουθούμε λοιπόν τη δική μας σχετική βιομηχανία. Γι' αυτό έχουμε επιφυλάξει σχετικά με την τροπολογία 96. Ενώ ε, συμφωνούμε με την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, ε, έχουμε ε, ανησυχίες σχετικά με την μείωση των ποσοτήτων των ζωοτροφών στην υδατοκαλλιέργεια. Με ενδιαφέρον άκουσα την τροπολογία 4 και την ε, αναφορά που κάνει στην ε, μέγιστη οικονομική βιώσιμη απόδοση. Θα ήθελα πολύ ε, να μάθω τι σχέση έχει αυτή με την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Όσον αφορά το θέμα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, γενικά συμφωνούμε με τις προτάσεις. Επιμένουμε όμως ε, ότι η κοινή αλλιευτική πολιτική θα πρέπει να πετύχει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015, ε, λαμβάνοντας υπόψη και το πολύπλοκο θέμα των ε, μικρών αλλιευμάτων. Θα πρέπει να συζητηθεί όμως εάν μπορούμε πράγματι να πετύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2015. Όσον αφορά τα, τις που είναι το αγαπημένο θέμα πολλών αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να ε, σταματήσει η απόρριψη ε, όχι μόνο των εμπορικών ειδών αλλά όλων των ειδών εκτός εάν είναι ε, ψάρια τα οποία έχουν δυνατότητα να επιβιώσουν μετά την απόρριψη τους στη θάλασσα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει η συμπεριφορά ε, πολλών ε, στην Αλία. Όσον αφορά τι μεταβάσιμε αλλιευτικέ ποσοστώσει, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τι διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη σε προαιρετική βάση για να ρυθμίσουν τι εθνικέ προτεραιότητε του. Το τελευταίο που θέλουμε είναι οι αλλιευτικέ ποσοστώσει να καταλήξουν στα χέρια μια ή δύο αλληλευτικών εκμεταλλεύσεων. Ε, επίσης ε, θα πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο ε, για να αναπτύξουν σχέδια διαχείρισης. Και θα ήθελα να πω ότι και η κύριος μα μας θα χαρεί πολύ να συνεργαστεί με τον Κρίς για να πετύχουμε τους στόχου αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Μάρτιν Κέλλερμαν και... Η συνάδελφο Φεραίρα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προλαλήσαντες εντόπισαν μερικά από τα πιο επίμαχα και κρίσιμα σημεία της έκθεσης και της αναθεώρησης της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Ο συνάδελφος Ντέιβιντ ε, στην αγνομοδότησή του ήταν πολύ εκτενής και διεξοδικός. Ε, είναι πραγματικά μεγάλη ποικιλομορφία στην αλληλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά την ε, σύσταση των ε, αλληλευτικών στόλων, τα χαρακτηριστικά τους, ε, τα αλληλευτικά εργαλεία, τα δίχτυα που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση των αλληλευτικών πόρων, όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά στα κράτη-μέλη. Οπότε μια κοινή ελευθερική πολιτική θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την ποικιλομορφία και την πολυμορφία. Μια πολιτική που θα διαφορεί για την διαφορετικότητα αυτή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν αυτή την πολυμορφία και ποικιλομορφία των καταστάσεων, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε μια διαχείριση σε τοπικό επίπεδο που θα αναμειγνύει τον κλάδο, τη παράκτιες ε, κοινότητες, όχι μόνο στην φάση της εφαρμογής της πολιτικής, αλλά και στη φάση της διαμόρφωσης, της χάρας χάραξη πολιτικής. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας είναι από τα πιο αρνητικά χαρακτηριστικά τη κοινή ελευθερική πολιτική μα σήμερα. Έχουμε μια κεντρική διαχείριση που δεν λαμβάνει υπόψη τοπικέ ιδιαιτερότητε και όταν εφαρμόζεται επί τόπου διαφέρει τελείω από περιοχή σε περιοχή. Οπότε τι περισσότερε φορέ ή δεν εφαρμόζεται καθόλου είτε έχει τα διαφορετικά, από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μερικέ φορέ και αντίθετα από τα αναμενόμενα και ζητωμένα αποτελέσματα. Και δυστυχώς η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, συνεχίζει αυτή την ε, πρόταση του συγκεντρωτισμού και της κεντρικής διαχείρισης. Γιατί το κεφάλαιο της περιφερειοποίησης και της αποκέντρωσης είναι πολύ ατελές και περιορισμένο. Επίσης έχουμε και κάποια νομικά κριτήρια και κάποιους τεχνικούς περιορισμούς αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέποτε δεν ήταν τα νομικά επιχειρήματα αρκετό λόγος για συγκεκριμένη κατεύθυνση των πολιτικών όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Δείτε τι συμβαίνει με το σύμφωνο που θα υπογράψει το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν ότι δεν είναι πρόσχημα αρκετή δικαιολογία τα νομικά προσκόμματα είναι σημαντικό να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην περιφερειοποίηση, στην αποκεντρωμένη διαχείριση. Επίση, όταν θέλουμε να μεταμορφώσουμε μια πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να τη γνωρίζουμε. Μία από τι σημαντικέ ελλείψει τη σημερινή ε, αλληλευτική πολιτική είναι ότι σε μεγάλο βαθμό είναι άγνωστη αυτή η πραγματικότητα. Η γνώση τη πραγματικότητα είναι πολύ μερική και ατελή. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για, την, για το πλεονάζον δυναμικό ε, δεν αρκεί να μιλάμε για την ε, υπερβολική αλληλευτική δυνατότητα. Θα πρέπει να δούμε σε ποια σκάφη, σε ποιους αλληλευτικούς στόλους, σε ποια κρατημέλη. Δεν ε, αρκεί να μιλάμε για πλεονάζοντα δυναμικό, θα πρέπει να δούμε πού εντοπίζεται θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει στοιχεία που να αποδεικνύουν γιατί κλάσματα, γιατί τμήματα του αλληλευτικού στόλου, γιατί αλληλευτικά αποθέματα και για ποια κράτη ισχύει αυτή η υπερβάλλουσα αλληλευτική δυνατότητα και η υπερβάλλουσα αλληλευτική προσπάθεια. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, πολύ πιο μεγάλη συγκεκριμενοποίηση για να διαμορφώσουμε σαφή αντίληψη για τη χρήση των συγκεκριμένων δικτυών, εργαλείων, ε, τα χαρακτηριστικά των αλευτικών στόλων και των αποθεμάτων. Αλλιώς ε, δεν θα καταλήξουμε σε καμία βελτίωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, μεταβιβάσιμες αλληλευτικές άδειες. Μερικοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στο θέμα αυτό. Σήμερα, ας είμαστε σοβαροί, επιστημονικές μελέτες που έχουμε μέχρι σήμερα για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων ε, καταλήγουν σε αντιφατικά αποτελέσματα. Ναι, μεν είχαμε θετικά αποτελέσματα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε άλλες περιπτώσεις είχαμε και αρνητικά αποτελέσματα. Και σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και ολέθρια αποτελέσματα από την εφαρμογή των μεταβιβασιμών αδειών. Νομίζω ότι καλύτερα να αφήσουμε στα κράτη-μέλη την απόφαση για το αν θέλουν να εφαρμόσουν ή όχι τέτοιο, τέτοιο σύστημα γιατί η εφαρμογή του συστήματος αυτού στις συγκεκριμένες πραγματικότητες, εκεί για παράδειγμα που υπάρχει η ε, υπεροχή της παράκτιας αλίας, ε, της αλίας μικρής ε, κλίμακας και της βιοτεχνικής αλίας, μπορεί τα αποτελέσματα να είναι ολέθρια, να επιβάλλουμε να εξαναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ένα καθεστώς διαχείρισης που η εμπειρία μας λέει ότι δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα και να εφαρμόσουμε για 15 χρόνια αυτό τον αναγκαστικό χαρακτήρα είναι κατά τη γνώμη μου παράλογο. Η εμπειρία μας έχει δείξει από την εφαρμογή των μετεβάσεων αλληλευτικών αδειών ότι έχουμε μείωση του αριθμού των σκαφών, αλλά αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη και μείωση της αλληλευτικής προσπάθειας. Αναφέρθηκε σε αυτό ο συνάδελφος Έκχοτ, Και μάλιστα, όταν μιλούμε για πλεονάζον δυναμικό, δεν αρκεί να μιλούμε μόνο για ποσότητα του ελευτικού στόλου. Θα πρέπει να μιλούμε και για ποιότητα, γιατί μείωση των ελευτικών σκαφών δεν σημαίνει αυτόματα και κατά ανάγκη μείωση τη ελευτικής προσπάθεια. Αντίθετα, αυτοί που απομένουν μετά τη μείωση των σκαφών είναι ικανοί για πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο εντατική ελευτική προσπάθεια. Με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην έχουμε μείωση της ε, αλίας, αλλά μπορεί να έχουμε και αύξηση της ε, αλίας. Άρα κανένα θετικό αποτέλεσμα για τη διαφύλαξη των αλευτικών αποθεμάτων. Ένας λόγος λοιπόν επιπλέον για να μην ε, επιβάλλουμε αυτό το σύστημα στα κράτη-μέλη, να μην έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Εναλλακτικέ λύσει υπάρχουν πολλές και διάφορες. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν υποβάλει πολλές τέτοιε εναλλακτικέ προτάσεις. Είναι σημαντικό και λαμβάνοντα υπόψη και το στοιχείο ποιότητα του στόλου, να δώσουμε έμφαση στην παράκτη αλία, βιοτεχνική αλία, αλία μικρής κλίμακας, που είναι πολύ πιο σημαντική για την αηφόρο ανάπτυξη της Έχουμε μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, που δυστυχώς δεν τα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια θετική διάκριση υπέρ της βιοτεχνικής μικρής κλίμακος αλίας. Γιατί εκεί η επιλεκτικότητα των αλληλευτικών εργαλείων είναι πολύ μεγαλύτερη. Η χρήση της ενέργειας είναι πολύ πιο ερθολογική και το δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης πολύ μεγαλύτερο. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να προταθεί διαφοροποιημένο καθεστώς για την βιοτεχνική αλληλεία, κάτι που δυστυχώς δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τοπική διαφοροποίηση ανάλογα με τα είδη των αλληλευτικών σκαφών για ορισμένα τμήματα των αλληλευτικών στόλων που είναι πιο βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη. Θα πρέπει να γίνουν τέτοιες διαφοροποίησεις και να λάβουμε υπόψη και την θετική εμπειρία από τη διαχείριση ε, των δύο μιλίων ε, σε ό,τι αφορά τις ε, ζώνες αποκλειστικής οικονομικής χρήσης. Δυστυχώ, τέτοιου είδου μέτρα δεν προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κακώ κατά τη γνώμη μου θα πρέπει στο μέλλον να ληφθούν υπόψη. Και τέλο. σε ό,τι αφορά τη σημασία που έχει καλύτερη διαμόρφωση γνώμης για την κατάσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων. Σήμερα έχουμε μια κοινή αλληλευτική πολιτική. Σε μεγάλο όμως βαθμό το κόστος της πολιτικής αυτής επιρρύπτεται στο, στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι λογικό. Δεν μπορούμε δηλαδή από τη μια να ζητούμε μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αλληλευτικών πόρων, μια και έχουμε κοινή αλληλευτική πολιτική, και να την ε, διαμορφώνουμε σε κεντρικό επίπεδο, αλλά να πληρώνουν τα σπασμένα, να πληρώνουν την ύφη μάλλον, τα κράτη-μέλη. Ακόμη και το κόστος για την απόκτηση των στοιχείων. Γιατί κάτι τέτοιο έχει ως συνέπεια αυτό που βλέπουμε σήμερα, ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει τεράστια ανεπάρκεια στοιχείων και γνώσης αντίληψης της κατάστασης των αλληλευτικών αποθεμάτων και των αλληλευτικών πόρων. Είναι λυπή τα στοιχεία που έχουμε και ο δημοσιονομικός κανονισμός των μέτρων της ΚΑΠ που ισχύει σήμερα προηγείται ακόμη και τις ε, τελευταίες συνθήκες. Είναι πολύ πιο παλιός. Οπότε θα πρέπει να αυξηθούν τα ποσοστά κοινοτικής χρηματοδότησης ε, για την ε, συγκέντρωση δεδομένων, κάτι που δεν γίνεται μέχρι στιγμής. Όλη την ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων την λαμβάνουν τα κράτη-μέλη, κακώς. Αυτά και είναι ένα θέμα που το αναφέρει ο κύριος Κριστέιβης στην έκθεση του. Τελευταίο σχόλιο. Μία κοινή ελευτική πολιτική θα πρέπει να έχει τρεις άρρηκτα συνδεδεμένες διαστάσεις. Την περιβαλλοντική, που είναι σημαντική, αλλά έχει και μία οικονομική και μία κοινωνική διάσταση ελευθερική πολιτική. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί την κοινωνική διάσταση. Ακόμη και η περιβαλλοντική διάσταση διακυβεύεται όταν διαφορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κοινωνική και κοινωνική διάσταση. Μας ανέφερε ο κύριος Στέβης στην περίπτωση των νησών Σέτλαντ. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε ε, πάλι φαινόμενα αλλιέων που μέσα στο χειμώνα και με κακοκαιρία για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Και όταν φτάσει σε αυτό το σημείο ο ψαράς να βγαίνει δηλαδή στη θάλασσα σε κακές συνθήκες μόνο και μόνο επειδή από αυτό εξαρτάται η επιβίωση οικογένειά του σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, τον ενδιαφέρει μόνο η επιβίωσή του. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την οικονομική πτυχή και την κοινωνική διάσταση. Γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα δίκαιο εισόδημα στους αλείς για να επιβιώσουν. Αλλιώς θα είναι δύσκολο να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε άλλο ε, και περιβαλλοντικό στόχο τη ελεύθερη πολιτική. Μπορούμε στα χαρτιά να έχουμε την καταπληκτικότερη νομοθεσία, αλλά θα παραμείνει μια νομοθεσία στα χαρτιά. Πολλέ φορέ καταβάλαμε προσπάθειε ελέγχου, αλλά αν ε, δεν βελτιώσουμε τον τρόπο ελέγχου, δυστυχώ οι προσπάθειε μα θα μείνουν ανεπαρκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερέιρα. Ακούσαμε όλους ε, τους σκιώδες εισηγητές. Ε, δεν κοίταξα το ρολόι, τους άφησα να μιλήσουν όσο θέλουν. Θα ήθελα να προτείνω ώστε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και για να μπορεί ε, και ο Κρις ε, να απαντήσει ως εισηγητής και να δώσουμε και το λόγο στην Κομισιόν να περιορίσουμε τον ε, χρόνο ομιλίας σε δύο λεπτά. Καταρχήν ο Πίτερ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την προσέγγιση της Επιτροπής και με την προσέγγιση ε, του εισηγητή. Θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την ε, αλλιευτική πολιτική, διότι πολλά ψάρια, υπερβολικά πολλά ψάρια αλλιεύονται από υπερβολικά πολλά σκάφη και υπερβολικά πολλά σκάφη, ε, ψάρια απορρίπτονται. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω κάποια ιδιαίτερα σημεία. Καταρχήν, μπορούμε να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι όσον αφορά τις ε, ε, μεθόδους της φιλικής προς το περιβάλλον. Ο εισηγητής ε, μιλάει για περισσότερα επιλεκτικά εργαλεία και φιλικά προς το περιβάλλον. Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι μέθοδοι που προστατεύουν το περιβάλλον η μέθοδοι και που δίνουν ε, ε, ε, στα ψάρια μια ευκαιρία να αποκατασταθούν, αναφέρονται υπερβολικά θολά και αόριστα εδώ. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Η αλλιευτική πολιτική αποτελεί αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων ε, δεν ε, δίδεται αρκετή σημασία στο, στις επιστημονικές εκθέσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει οι επιστημονικές εκθέσεις να ε, λάβουν περισσότερη σημασία και να το αναφέρουμε αυτό περισσότερο στην έκθεση. Δεύτερον, οι φορολαφρύνσεις για τους αλίες που εγκαταλείπουν την ε, αλία. Στη χώρα μου υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αποχωρούν από την αλία, κάτι το οποίο ε, συμβάλλει στην μείωση του υπερβολικού αλλιευτικού στόλου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, κατά τα πρώτα χρόνια της νέας σταδιοδρομίας τους με φορολαφρύνσεις, για παράδειγμα, διότι έτσι συμβάλλουν στη μείωση της αλληλευτικής ικανότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα. Και όσον αφορά τη δική μας ε, συμπεριφορά, όταν ε, πηγαίνω στο Στρασβούργο και περνάω από εστιατόρια Σούση, βλέπω το μισό κοινοβούλιο εκεί μέσα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τη δική μας ε, συμπεριφορά. Και ένα διαδικαστικό. Ε, στην... Ε, σας παρακαλώ μην το υπολογίσετε αυτό στο χρόνο ε, ομιλίας μου. Ε, ήθελα να μιλήσω για τον... Ε, θα ήθελα να μιλήσω για τον χρόνο ομιλίας με... Μου κάνει εντύπωση που περιορίζεται το χρόνο για τον ε, δεύτερο γύρο των ομιλητών, ε, ενώ δεν το περιορίζεται για το πρώτο. Δεν θα πρέπει να το ε, συζητήσουν αυτό οι συντονιστές. Είναι σημαντικό θέμα, είναι σαφές αυτό. Ε, μπορώ να σας πω όμως ότι για τους εισηγητές ε, όλα τα θέματα είναι σημαντικά. Ε, ο καθένας θέλει για το θέμα του περισσότερο χρόνο. Δώσαμε, προβλέψαμε λοιπόν λίγο περισσότερο χρόνο για το θέμα αυτό. Und Laios Ja, So, dann fangen wir an mit Jonas. Ξεκινάμε με τον Γιάννος, παρακαλώ. Ε, köszönöm a szót, elnök úr. Ε, valóban nem Jónás, hanem János. Ez két, két különböző név. Nos, tisztelt kollégák! Ευχαριστώ ε, πολύ κύριε Πρόεδρε. Γιάννος είναι το όνομά μου και όχι Γιώνας, είναι διαφορετικά ονόματα αυτά. Άκουσα με προσοχή Ε, ο κάθε ομιλητής όμως, όλοι οι ομιλητές μίλησαν για ε, την αλία στη θάλασσα και όχι την αλία ε, στα γλυκά νερά. Το 75% των αλλιέων αλλιεύουν στη θάλασσα και το 1 τέταρτο στα γλυκά νερά. Και Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντική η προστασία των ε, ε, αλλιευμάτων, των αποθεμάτων ε, στη θάλασσα είναι πολύ σημαντική, αλλά επίσης σημαντική είναι και η αποκατάσταση των αλλιευμάτων, των αποθεμάτων στα εσωτερικά ύδατα, στον Δούναβη και σε άλλα ποτάμια. Πολλοί αναφέρθηκαν στο Σολομό. Πόσο νόστιμο είναι το ψάρι αυτό. Έχετε ε, φάει όμως και κυπρίνουσα ή πέστροφα από το Δούναβι. Εγώ θα ήθελα να σας προτείνω να φάτε και αυτά τα ψάρια και θα δείτε ότι είναι εξίσου νόστιμα ψάρια με τα θαλάσσια είδη. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Chris Davis να ανακαλέσει όλες ε, τις τροπολογίες που είναι εις βάρος των ε, ηχθείων ε, των ε, γλυκών υδάτων και αν δεν το κάνει θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να μην στηρίξουν τις τροπολογίες αυτές διότι βρίσκω ότι προκαλούν διακρίσεις και ότι δεν είναι επικοδομητικές και στο, στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει αλία των γλυκών υδάτων και Ε, θα πρέπει άλλωστε να απολογηθείτε απέναντι και στους ε, Βρετανούς αλλιέους ε, που εκτρέφουν πέστροφα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη βιοπικιλότητα και στα γλυκά ύδατα. Κύριε Ντέιβι, σας παρακαλώ να ανακαλέσετε τις σχετικές προτάσεις. ευχαριστώ ο Καλ Σλούτερ και κατόπιν ο Ρίχαρτ Σίπερ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ, Κρίση, για την έκθεση. Ο, ο τίτλος όμως πιστεύω ότι είναι λάθος. Δεν θα έπρεπε να είναι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠΑ, αλλά η μεταρρύθμιση της ε, διαχείρισης της θάλασσας. Εμείς θα έπρεπε να στείλουμε την κρίση στο Συμβούλιο για τις διαπραγματεύσεις για τις ε, άδειες. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι αυτές οι μεταβάσιμες άδειες. Η κανονική αγορά είναι ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αυτή, εγώ έτσι το έχω αναλύσει. Αλλά μπορώ να πω τότε ναι μόνο υπό, μια, υπό έναν όρο, διότι ανέφερε ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα ψάρια να έχουν σεξουαλικές επαφές. Αν και στη Σουηδία μπορεί να έχει άλλες, ε, ε, άλλα νοήματα, γιατί όταν πας σε μια πόρνη λέει ότι πας και τρως ε, μπακαλιάρο. Οπότε καταλαβαίνεις μπορεί να παρεξηγηθούμε στη Σουηδία. Μας περιπτώσει ε, το λογικό συμπέρασμα είναι ότι οι άδειε και οι ποσοστώσει θα πρέπει να γίνονται, δίνονται σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Και αν ένα επαγγελματία αλλιέα θέλει να αλλιέψει θα πρέπει να αγοράσει την ποσόστοση αυτή από τον κάθε πολίτη. Τότε θα είχαμε αλληλευτική πολιτική που θα ήταν δυνατόν να τη διαχειριστούμε, νομίζω. Ακόμα και αν τεχνικά είναι περίπλοκο, πιστεύω ότι αυτή η ιδέα ότι τα ψάρια ανήκουν σε κάθε μονομένο πολίτη είναι καλή και είναι λάθο να δίνουμε τι ποσοστώσει στα μεγαλύτερα σκάφη και ούτω καθεξής. Η λογική θα έπρεπε να είναι ότι ο κάθε ένας πολίτης έχει ένα δικαίωμα και αν θες να τα χρησιμοποιήσεις πρέπει να τα αγοράσει. Γιατί είναι κοινό πόρος. Οι αλληλεί δεν βάλαν τα ψάρια στη θάλασσα, απλώς εκμεταλλεύονται ένα φυσικό πόρο. Επίτα από την περασμένη χρονιά ήμουν εισηγητής για την, απο, για την απόρριψη των ε, περισσευούμενων αλλιευμάτων. Είναι πραγματικά σημαντικό να μην δημιουργήσουμε κρυφή αγορά ή δεύτερη αγορά για τις απορρίψεις. Θα πρέπει κανείς να πληρώνεται μόνο για το πραγματικό κόστος που επιφέρει η... το να φέρει κανείς αυτά τα ψάρια προς απόρριψη στο λιμάνι. Τώρα για την καλλιέργεια, τις σα συμφωνώ με τη βιωσιμότητα, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή στα χορτοφάγα ψάρια. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα μας, έβλεπε, θα μας ε, βοηθούσε να αποφύγουμε το πρόβλημα της απόρριψης και των ε, παραλιευμάτων κτλ. Θα ήταν χρήσιμο να το εστιάσουμε σε αυτό. Είναι μια μεταρρύθμιση λοιπόν της διαχείρισης της θάλασσας και θα πρέπει να ασχολούνται με αυτήν μόνο οι άνθρωποι της Επιτροπής Αλίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζήπερ. Ευχαριστώ, Καρλ Σλίτερ, ο Ρίχαρτ Ζήπερ. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και του κοιόδη εισηγητέ ε, για τη δουλειά που έχει γίνει. Ε, είναι σαφέ ότι μιλάμε για έναν φυσικό πόρο και για μια ευθύνη την οποία πρέπει να αναλάβουμε από κοινού. Και στην Ευρώπη δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στο θέμα αυτό το δείχνουν αυτό τα στοιχεία. Κάθε τέταρτο ψάρι απορρίπτεται πάλι στη θάλασσα και μάλιστα νεκρό και το 60% των καταναλώνων ψαριών προέρχεται από ε, ε, εισαγωγές. Στην ε, πρώτη παράγραφο της αιτιολογικής σκέψης του Chris Davis ε, τα γράφει αυτά. Οι προτάσεις πηγαίνουν απολύτως προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την, ε, τα, τα δεδομένα που υπάρχουν και να μην μιλάμε μόνο για γνώμες ε, και απόψεις, αλλά να γνωρίζουμε περί τίνος μιλάμε και επίσης να κατανείμουμε τους ρόλους σωστά ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, και τα θεσμικά όργανα. Ε, θα πρέπει να αφήσουμε στα κράτη-μέλη την μικροδιαχείριση ταυτόχρονα για την βιοτεχνική αλληλεία, για την αλληλεία μικρής κλίμακας θα πρέπει να προβλέψουμε και ε, σχετική ποσόστοση. Ε, δεν θα πρέπει όμως ε, η κοινότητα να παρεμβαίνει σε αυτήν την μικροδιαχείριση. Ταυτόχρονα θέλουμε υψηλό βαθμό διαφάνειας, διότι δεν υπάρχει διαφάνεια στον τομέα αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφή τα στοιχεία. Ε, εάν ε, είχαμε ε, σαφέστερα στοιχεία δεν θα υπήρχε ναι, αυτές οι ζημιές πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερε ο, ε, ο Και επίσης θα πρέπει οι κυρώσεις να είναι επαρκείς και σκληρές ώστε να αποτρέπουμε ε, κακές πρακτικές. Ε, χαίρομαι που η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, μπορεί ε, να πει τη γνώμη τη για το θέμα αυτό. Τώρα αφήσουμε τέτοια θέματα αποκλειστικά στα χέρια των Ελλήνων πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίπερ. Ο Πόκρο Λάιο έχει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Uh, Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ προέρχομαι από μια χώρα που δεν έχει ε, πρόσβαση στη θάλασσα και γι' αυτό και δεν θα μιλήσω πολύ για την θάλασσα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ε, τομείς όπου αυτή η έκθεση μπορεί να αναβαθμιστεί. Ένας ε, τομέας λείπει, η χρηματοδότηση. Έχουμε μόνο μια πρόταση. Στο ολόκληρο το σύντομα λογικό σημείωμα που μιλά για τη χρηματοδότηση και λέει στην πρώτη παράγραφο ότι η ελευθερική βιομηχανία είναι πολύ κερδοφόρα και ότι ε, μπορεί να αναζωογονηθεί μόνο με επιδοτήσεις. Αν αυτό το τοποθετήσουμε στο ευρύτερο πλαίσιο, θα δεις γιατί υπάρχει παρακμή της ευρωπαϊκής δύναμης. Πολλά χρήματα δαπανώνται για κάτι το οποίο είναι πλήρης σπατάλη. Κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων. Οι επιδοτήσει μπορούν να αιτιολογηθούν αν είναι προσωρινές, προσωρινά μέτρα για να χρηματοδοτήσουν την εξάλληψη ας πούμε της υπερβολ... του... μεγάλου στόλου των υπερβολ... της υπερβολικής δυνατότητας. Εδώ χρησιμοποιούμε τις επιδοτήσεις για να διατηρήσουμε αυτόν τον μεγάλο στόλο, πράγμα που είναι αρνητικό. Εγώ ήμουν μέλος της Επιτροπής Προπολογισμού μέχρι πρόσφατα και ξέρω πόσα χρήματα δαπανώνται για πράγματα που ω συνέπεια δεν παράγουν καμιά θετική αξία. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε έναν συντονισμό και συνεργασία με την Επιτροπή Αλληλείας και με την Επιτροπή Προϋπολογισμού, γιατί αν αναλύσει κανείς τις τροπολογίες δεν, υπάρχει, δεν έχει νόημα Χωρίς να έχουμε βιώσιμη ε, χρηματοδότηση, ε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και βιώσιμη αλία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν για πέντε λεπτά. Ερνέστο Λάτο από την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, παρακαλώ. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, let me start... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κομισιόν υποστηρίζει και είναι ευτυχής με την έκθεση που επέβαλε ο εισηγητής Ντέιβις. Εν γέννη, συμμεριζόμαστε ε, τις απόψεις του και καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση που ενισχύει τη δική μας άποψη υπέρ της ε, μεταρρύθμισης της πολιτικής. Εν γέννη λοιπόν συμφωνούμε με την πρόταση αυτή. Δεν θα σχολιάσω μεμονωμένα τις τροπολογίες, αλλά κάποιες από τις πιο σημαντικές, που, μάλλον από, θα σχολιάσω κάποια εδάφια της αιτιολογικής σκέψης ε, του εισηγητή. Εμείς καλωσορίζουμε κάθε πρωτοβουλία για αποκατάσταση των ύφθη αποθεμάτων. Αυτό έχουμε πει, δεν υπάρχει η κυριαρχία των περιβαλλοντικών στόχων στο άρθρο 39 της συνθήκης, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι μόνο ευνοώντα του περιβαλλοντικού στόχου μπορούμε στην πράξη να επιτύχουμε ισορροπημένους στόχους για την ΚΑΛΠ στο πλαίσιο του άρθρου 39 της συνθήκης. Άρα λοιπόν ανάκτηση των νυχθεί αποθεμάτων είναι προϋπόθεση για τους ισορροπημένους στόχους της ΚΑΛΠ και την επίτευξη αυτών. Έπειτα για το θέμα της, ε, των ε, σχεδίων διαχείρισης είναι σημαντικό όταν ορίζονται τα ετήσια τάκ να ορίζονται με τρόπο ώστε οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη ε, προγράμματα διαχείρισης να τηρούνται. Πρέπει αυτό να το κάνουμε με τρόπο που να σεβόμαστε την αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου ε, για την θέσπιση των, αιτιαίων δυνατο... των συγγνώμη, ετησίων δυνατοτήτων αλήψης σύμφωνα με το άρθρο 43.3 να υπάρξει μεν κάποια πειθαρχία αλλά που θα τηρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 43.3 όσον αφορά την απαγόρευση της ε, δε συμφωνούμε φυσικά ε, και ευχαριστούμε τον κύριο Τέβης που υποστηρίζει την άποψή μας. Πιστεύω, Πρόεδρε, ότι για να απαμβλύνουμε τις αμφιβολίες για αυτή την πρόταση υπόθηκε και σήμερα το πρωί αυτό εξάλλου ότι η πρότασή μας για να καταστήσουμε υποχρεωτική την εκφόρτωση όλων των αλλιευμάτων ε, ορισμένων ειδών Ακόμα και για τα μικρά ψάρια, αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία αγοράς για τα μικρά ψάρια. Αυτό υπόθηκε ως αντίρρηση. Αυτό όμως δεν είναι η πρόθεσή μας. Ενώ θα κάνουμε αυτή την πρόταση, συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να εξασφαλίσουμε την ελαχιστοποίηση το της αλίευσης των μικρών νεαρών ψαριών. Μέσω της βελτίωσης της αλληλευτικής δραστηριότητας από την, με βάση την νομοθεσία αλλά και δίνοντας οικονομικά κίνητρα στην επιλογή της ε, επιλεκτικής αλληλείας. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν όλο αυτό. Θα φτιάξουμε μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η επιλεξιμότητα, μάλλον η επιλεκτικότητα της αλληλευτικής δραστηριότητας ε, καταρχήν θα μειωθεί. Αλλά πείτε γνωρίζουμε πως θα λειτουργησει λοιπον ολο αυτο θα φτιαξουμε μετρα ωστε να εξασφαλισουμε οτι η μαλλον επιλεκτικοτητα της αλληλευτικης δραστηριοτητας καταρχην θα μειωθει αλλα πειτε γνωριζουμε πως αυτη στον πραγματικό κόσμο αυτή η μείωση δεν μπορεί να εκμηδενιστεί, δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Αναπόφευκτα λοιπόν, όση πρόοδο και αν κάνουμε για τη μείωση αυτής της δραστηριότητας, των παράπλευρων μάλλον ε, θα υπάρχει κάποιος αριθμός μικρών ψαριών και δεν θα μπορούμε να, τους αφήσουμε, να τα αφήσουμε στις προβλήτες, αλλά κάτι πρέπει να τα κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε τι θα τα κάνουμε αυτά τα ανεπιθύμητα ψάρια που πρέπει να εκφορτωθούν. Θα είναι ωστόσο πολύ μικρότερος ο όγκος από αυτό που γίνεται σήμερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και μπορώ μόνο να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο εισηγητή. Ότι πρέπει δηλαδή να υποδείξουμε ότι η πρόταση της Κομισιόν βασικά θα είναι να μπορούν τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν το εθνικό σύστημα για τι μεταβιβάσιμε ελευτικέ παραχωρήσεις με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν τις θεμητέ ανησυχίε που εκφράζονται για πιθανή σώρευση ή για πιθανού τομεί ή τμήματα τα οποία εξαιρούνται από δικαιώματα, λευτικά δικαιώματα. Εδώ έχουμε εμπειρίες από διάφορες χώρες του κόσμου, στη ΣΥΠΑ και στην Ένωση βέβαια και φυσικά η Κομισιόν ποτέ δεν θα πει ότι ε, είναι το τέλειο σύστημα οι τι ε, παραχωρήσεις και ότι λύνουν το πρόβλημα, αλλά σίγουρα το λύνει πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλη εναλλακτική που έχουμε στη διάθεσή μας. Η εμπειρία μας ε, είναι ότι όταν δεν προστατεύεται κάποιο μάλλον κάποια παράκτια αλλιευτική κοινότητα είναι διότι η, προ... η αλληλευτική πολιτική, το σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί κατά αυτόν τον τρόπο, όπως στην Ισλανδία. Όμως, όταν τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να προστατεύσουν τις τη μικρή κλίμακα ε, αλληλεία, ή τις ε, τοπικές παράκτιες κοινωνικές κοινότητες όπως στη Νέα Ζηλανδία, στη ΣΥΠΑ έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα, παραδείγματα από τη Χιλή το επιτυχάνουν. Όλα εξαρτούνται από το σχεδιασμό της πολιτικής. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ως μοιραίο το σύστημα των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων. Τίποτα δεν είναι αναπόφευκτο. Τα πάντα εξαρτούνται από το σχεδιασμό. Και ο σχεδιασμός στη δική μας πρόταση έχει ε, γίνει ο σχεδιασμός με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται περιθώριο λιγμού στα ίδια τα κρατημέλη. Για τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για αλληλεία μικρής κλίμακας και μάλιστα θα χρησιμοποιήσω και μια φράση που χρησιμοποιήθηκε εδώ τη δυνατότητα δηλαδή δημιουργία ενό συστήματο με καταχωνομή ποσοστώσεων ανάμεσα στα κάτι που θα ανταμείβει όσου ε, κάνουν το σωστό. Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά θα σα θυμίσω, όπω είπε και ο κύριο Ντέβι ο ίδιο, ότι σήμερα αυτή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το ζήτημα είναι λοιπόν ως εσείς ως συνομοθέτες, αν πιστεύετε πως δεν θα πρέπει να είναι μόνο α, α, απόλυτα ελεύθερα τα κρατη να κάνουν αυτό που θέλουν. Θα πρέπει να έχουν κάποιο είδος γενική υποχρέωση υπό το εθνικό του σύστημα, ας πούμε, να θεσπίζουν προτεραιότητες ή συστήματα κατανομής των αληφτικών δικαιωμάτων που θα ευνοήσουν περισσότερο την μικρή κλίμακα αλληλεία ή τη βιώσιμη πρακτική αλληλεία. Φυσικά όλα αυτά θα τα εξετάσουμε με ευνοϊκό Ευνοϊκή διάθεση. Αυτή τη στιγμή είναι αρμοδιότητα κρατών μελών, αποκλειστικότητα. Ε, τώρα, αν θα πρέπει να παραμείνει αποκλειστικότητα ή όχι είναι το θέμα. Και το θέμα τώρα τη της επιμένουμε ότι θέλουμε να ευνοήσουμε τις ιδετοκαλλιέργειε απόλυτα όμως συμβατές με τον σεβασμό του περιβαλλοντικού δικαίου στην Ένωση. Και ένα θέμα που αφορά τις ζωοτροφέ και καταλαβαίνω την νόημα των προτάσεων του εισηγητή. Το θέμα όμως είναι ότι η παγκοσμιοποιημένη αγορά για τις ε, τροφές για τα ψάρια είναι τέτοια που δεν είναι εύκολο να κάνουμε καλό υπολογισμό και να συγκρίνουμε τις υδατοκαλλιέργειες με τις τροφές για τα ψάρια. Προέρχονται αυτές από τη Χιλή και από το Περού που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο να υπάρξει λοιπόν σαφής ε, συσχετισμός εκεί. Για το θέμα της διαφάνειας φυσικά και συμφωνούμε. Όσο πιο διαφανές είναι το σύστημα τόσο καλύτερο για τα λιγοστά ερωτήματα όσον αφορά την περιφερειοποίηση. Περιφερειοποίηση και κατά πόσο θα πρέπει πιο λεπτομερώς να νομοθετήσουμε από ό,τι σε αυτή την πρόταση, νομίζω πως είναι πολύ εύκολο για μένα και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι οι νομικοί δεν μας αφήνουν να το κάνουμε αυτό. Είναι ένας τομέας όπου η συνθήκη δεν ε, έχει δεν περιλαμβάνει καμιά πρόβλεψη για την λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο να νομοθετήσει κανείς σε τέτοια θέματα και για, περιφερειακά και γι' αυτό δεν το κάναμε. Και έχουμε όμως μια πιο ουσιαστική ερώτηση, ε, ένα θέμα πιο σημαντικό. Είναι καλή ιδέα. Εμείς την περιφερειακή λήψη αποφάσεων την βλέπουμε σε ένα θέμα που θα πρέπει να εξελιχθεί. Δεν έχουμε κάποιο κάποια μαγική συνταγή, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί μέσα στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει καθώς προχωράμε. Και θα ήταν ίσως λάθος να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε με πολλές λεπτομέρειες ε, πώς θα γίνει αυτή η περιφερειακή λήψη αποφάσεων, γιατί μπορεί να μην προσαρμόζεται σε διάφορες ε, περιστάσεις. Αντί λοιπόν να έχουμε ένα πολύ λεπτομερές προσχέδιο για το πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη, θα το βλέπουμε ως μια διαδικασία εκμάθησης όπου η πρακτική, η πράξη θα μας δείξει ε, πώς στην πορεία θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Για τις παράκτης ε, κοινότητες και τις επενδύσεις εκεί, ναι, όντως όταν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την πρόταση αυτή για την αλληλεία και το, ταμείο, το θαλάσσιο ταμείο, έχουμε προτείνει σημαντική αύξηση, μάλλον μετακίνηση από τα ταμεία που αφιερώνονται στη διάλυση σκαφών και εκείνα που τα κονδύλια τα οποία δεν δαπανώνται πια για την διάλυση πλοίων θα πάνε στην ανάπτυξη των παρακτήων αλλιευτικών περιοχών. Το Ταμείο λοιπόν Αλίες και Θαλάσσης θα μετακινήσει κονδύλια από την διάλυση σκαφών στην ε, ανάπτυξη των παρακτήων κοινοτήτων. Τώρα, δεν έχουμε πολύ τελευταίες πληροφορίες για τους εργαζόμενους, αν εκτιμούμε όμως ότι πρόκειται για 10% μίνιμουμ μη Ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται στα ευρωπαϊκά ελευτικά σκάφη. Δεν είναι τα τελευταία στοιχεία αυτά που όμως, αλλά η αναλογία αυτή φαίνεται τα τελευταία χρόνια να έχει αυξητική τάση. τα κράτη-μέλη θα υπογράψουν σύντομα την σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, είναι θέμα των κρατών μελών, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και ελπίζουμε ότι θα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις και για τους εργαζόμενους στη θάλασσα περισσότερα στοιχεία για να έχουμε ε, επιτυχή πολιτική. Συμφωνούμε και γι' αυτό. Να σας πω μόνο ότι δεν είναι ακριβές ότι πρόκειται για κοινή πολιτική, αλλά τα στοιχεία πρέπει να τα πληρώνουν. Τη συλλογή των στοιχείων την, πληρώνει τα κράτη, την πληρώνουν τα κατημέλη. Σήμερα 50% ε, χρηματοδοτεί η Ένωση για τη δαπάνη αυτή και στο πλαίσιο του Ταμείου Θαλάσσης ε, προτείνουμε 350 εκατομμύρια ευρώ για τη συλλογή των στοιχείων και με μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής της Ένωσης, μέχρι και 65% θα φτάνει αυτό του συνόλου της δαπάνης. Νομίζω πως έτσι απάντησα σε όλες σας τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις αυτές. Τελευταίος έχει το λόγο ο εισηγητής Κριστέιβης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα προσπαθήσω εν συντομία να ανακεφαλαιώσω. Όπω είπα, του τελευταίους μήνε παρακολούθησα πολλέ συνεδριάσει με εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ήταν πραγματικά επαρηλημμένε και ε, ήταν πραγματικά σαν καθαρτήριο για του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω η σημερινή συνεδρία να ήταν πιο ανακουφιστική Είμαι πολύ τυχερός που έχω τέτοιους σκιώδεις ηγητές για αυτή τη γνωμοδότηση και με την κυρία Ρόντος θα έχουμε την αρμόδια στην Αλληλευτική Επιτροπή, θα έχουμε αγαστή συνεργασία. Ήδη είπε ότι ευθυγραμμίζεται και η συγκήτρια που κάνει καταπληκτικό έργο με την κρατούσα γνώμη και στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να μιλήσω για ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τα ψάρια α, του γλυκού νερού δεν ήθελα να κάνω καμία διάκριση. Κύριε Φιέλνερ, η χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική, αλλά υπάρχει ξεχωριστό χρηματοδοτικός κανονισμός. Φαντάζομαι ότι δεν θα υποβάλλετε τέτοιες προτάσεις στη δική μου γνωμοδότηση. Τώρα, η Λίντα Μακάβαν μίλησε για τις απορρίψεις μεταξύ άλλων. Ρώτησε για εναλλακτικέ προτάσει και λύσει. Όντω, αυτό είπα και στι εισαγωγικέ μου παρατηρήσει. Η απαγόρευση των απορρίψεων δημιουργεί μια δυναμική. Δεν είναι μια στατική κατάσταση. Δημιουργεί μια δυναμική εξέλιξη. Και είπαμε ότι δεν υπήρχαν ε, επιλεκτικά ε, εργαλεία. Ε, με το που απαγορεύτηκε όμως σε μια χώρα η ε, η πολιτική των απορρίψεων, αμέσω εμφανίστηκαν επιλεκτικά αλληλευτικά εργαλεία. Το σύστημα των μεταβάσεων ελευτικών παραχωρήσεων στην ε, Ολλανδία δεν δημιούργησε πλεονάζο δυναμικό, είπε κάποιο. Δεν είναι ότι η αρχή έχει πρόβλημα. Το σύστημα είναι προβληματικό και θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε κάποιο είδου ε, ε, συστήματος μεταβιβάσιμων αλληλευτικών αδειών. Χρειάζεται και αυτό αλλαγή. Είπαμε ότι μέχρι το 2015 θα υλοποιηθεί ο στόχος. Βέβαια, η, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το SFMSY ε, για το πώς θα περιοριστεί η θνησιμότητα των ψαριών. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό για όλα τα ελευτικά είδη μέχρι το 2015, μέχρι το 2020. Εξαρτάται από τον ορισμό που θα ε, επιδιώξουμε. Σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ε, οικονομική απόδοση. Εγώ είπα ότι θέλω αποκατάσταση των ελευτικών αποθεμάτων στα επίπεδα της προηγούμενης ε, πεντα, Βέβαια είναι και θέμα ερμηνείας εδώ. Ποια είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ των αλληλευτικών στόχων και των αλληλευτικών στόχων, συγγνώμη, και της αποδοτικότητάς τους. Εκεί ίσως γίνουν κάποιες ε, τροποποίησεις. Η βασική μου διαφορά, οι βασικές μου διαφωνίες ε, έχω σχέση με τα σχόλια του κυρίου Φεραίρα, δεν θα σα εκπλήσει αυτό. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Κύριε Φεραίρα, είπατε ότι οι αλλοί μερικέ φορέ για να επιβιώσουν ε, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ναι, αλλά γιατί ακριβώς ε, είναι όλο και πιο δύσκολη η αλία, δεν υπάρχει πια εύκολα προσιτό ψάρι. Αυτό δείχνει πόσο, σε πόσο κακή κατάσταση βρίσκονται τα αλλιευτικά αποθέματα. Γι' αυτό και η προστασία τη παράκτη αλληλεία είναι ευθύνη των κρατών μελών, παρόλο που θα υπάρχουν, θα δοθούν και κονδύλια από τον αλληλευτικό κανονισμό. Αλλά δεν λέμε από τη μια μεριά να λέμε θέλουμε μεγαλύτερη περιφερειοποίηση και αποκέντρωση και από την άλλη να ζητούμε περισσότερα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόθεση της, της παράκτης αλίας, μικρή μικρής κλίμακος και βιοτεχνικής. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε για όλα τις Βρυξέλλες, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε τις επιδοτήσεις αλληλευτικών προσπαθειών που είναι, δεν είναι επικερδής. Αυτό όμως ουσιαστικά διονύζει μια κακή αλληλεία Τέλος, Κρίστοφερ Φιέλνερ, είπατε πολύ σωστά ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από ε, λίγο κόσμο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από λίγες κυβερνήσεις ουσιαστικά. Ε, μια μικρή ομάδα υπουργών αλίας. Και τελικά λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν βραχυπρόθεσμες αποφάσεις αντί να έχουν μια πιο διορατική και μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτό πιστεύω θα είναι το πιο σωστό μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε για καλύτερη και βιώσιμη διαχείριση αλίας προς τους αλίες. Το ίδιο ισχύει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτός είναι ο κίνδυνος, αυτός ο κίνδυνος ελοχεύει. Ένας μικρός αριθμός ευρωβουλευτών που είναι πιο εξοικειωμένοι με τα θέματα αυτά και έχουν κίνητρο να προστατεύσουν και τα εθνικά τους συμφέροντα, θα εμφανιστούν στις ομάδες εργασίας, ε, στο Κοινοβουλίο και εκεί που θα ληφθούν αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή, ενώ η πλειοψηφία θα πει ναι, είμαστε υπέρ τη αναθεώρηση τη ΚΑΠΑ, αλλά δεν είναι πρωταρχικό ζήτημα. Και θα πουσιάζουν εκεί που θα αποφασιστούν ε, οι πολιτικέ. Γιατί ε, η πολιτική καθορίζεται από αυτούς που λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να δώσουμε το παρόν. Ευχαριστώ Κριστέβης. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να συζητήσουμε εις βάθος το θέμα αυτό. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 9 Μαρτίου στις 12 η ώρα. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσουμε στις 12 Απριλίου και η έκθεση στην Επιτροπή Αλληλείας. Θα ε, ψηφιστεί στην Επιτροπή 10 Ιουλίου ε, και, στην, ε, και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. 25 Απριλίου λοιπόν θα είναι η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας, στην ΕΝΒΗ. Είναι σημαντική η έκθεση αυτή. Συνδέεται και με το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας, με την αλληλευτική πολιτική η αριφτική πολιτική και η γεωργική πολιτική μέχρι τώρα πάντα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευση και κλεισμένων των θυρών. Ενώ τώρα πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να γίνουν πιο διαφανείς οι πολιτικές αυτές. Οι σκιώδεις εισηγητές ε, και, και οι εισηγητές των δύο επιτροπών έχουν σημαντική ευθύνη και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό. Προτού να ε, προχωρήσω στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα ε, ε προσκεκλημένων από την Φινλανδία. Ε, είναι προσκεκλημένη της ε, Σάτου Χάση. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φτάνουμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης και... Το θέμα εδώ είναι η κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα των προϊόντων αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια. Η Εισηγητής είναι ο συνάδελφος Φερέιρα. 30 λεπτά έχουμε χρόνο για την έκθεση αυτή. Ε, θέλουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό γύρω στις 11 και μισή. Πρώτα έχει το λόγο εισηγητής ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ. Ο λόγο ύπαρξη αυτή τη έκθεση προκύπτει από το γεγονό ότι η οργάνωση ε, και ο συντονισμός των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας έχει άμεσες επιπτώσεις στην ε, βιωσιμότητα των αλλιευτικών πόρων και των θαλασσίων οικοσυστημάτων αλλά και στη δημόσια υγεία και την επισητιστική ασφάλεια των πληθυσμών. Με αυτές τις προτινόμενες τροπολογίες προσπαθώ να δώσω απάντηση σε αυτά τα δύο ζητήματα. Από τη μια πλευρά τα περιβαλλοντικά και από την άλλη τα θέματα δημόσιας υγείας και επισητιστικής ασφάλειας. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η περιβαλλοντική διάσταση είναι αλληλένδετη με την οικονομική και την κοινωνική στην περίπτωση της αλληλείας. Άρα λοιπόν, για να επιτύχουμε βελτίωση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και της αλληλείας, πρέπει να λάβουμε διάφορα μέτρα που να καλύπτουν το κοινωνικό και το οικονομικό πεδίο. Και αυτό είναι το γενικό όραμα το οποίο αιτιολογεί την ύπαρξη αυτής της έκθεσης. Είναι σημαντικό λοιπόν να αξιοποιηθεί ε, ο ρόλος της αλληλείας μικρής κλίμακας και της αλληλείας με παραδοσιακά μέσα, και να στηριχθούν οι παραγωγοί που ανήκουν σε αυτόν τον τομέα του στόλου. Και ε, το τομέας αυτός του στόλου σήμερα είναι πολύ περιορισμένα ενταγμένος στην κοινή οργάνωση των αγορών και επίσης αυτό είναι ορατό σε κάποια κράτη-μέλη και είναι σημαντικό να μην λησμονούμε ότι αυτοί οι τομείς Ε, είναι συνδεδεμένη με μια πιο συντηρητική εκμετάλλευση των πόρων, επειδή καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και επειδή οι αλληλευτικέ τεχνικέ που χρησιμοποιούν έχουν μεγαλύτερη επιλεκτικότητα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Ντέβι ότι ό,τι αφορά την μικρή αλληλεία, τη μικρή κλίμακα αλληλεία είναι, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αν και μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το επίπεδο για να βοηθήσουμε την μικρή κλίμακα αλληλεία. Εξάλλου, τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολο να υπάρχει αυτή η θετική ε, διάκριση υπέρ της μικρής κλίμακας αλίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν εδώ τι θα κάνουμε στο επίπεδο της κοινή οργάνωσης αγοράς. Κατά την γνώμη μου, η ΚΟΑ θα πρέπει να αυξήσει τη συμβολή της στην εξασφάλιση των εισοδημάτων του τομέα και στη βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων αλληλείας και δατοκαλλιέργειας, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Αυτό το ζήτημα είναι ε, αλληλένδετο με τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων που συντελεί στον καθορισμό της αλληλευτικής προσπάθειας σε επίπεδα συμβατά με την ε, ικανότητα αυτοανανέωσης των αλληλευτικών αποθεμάτων. Αυτή η θεώρηση δεν συμβιβάζεται με την εξάρθρωση των δημόσιων μέσων ρύθμισης των αγορών. Αντίθετος, χρειάζεται φιλόδοξη ενίσχυσή τους. Και με αυτό την πρόταση της Κομισιόν ε, αυτό θα πρέπει να γίνει. Μια ευφυής ενίσχυση τον ε, ΚΟΑ ώστε να δοθούν απαντήσεις στις βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλληλείς, δηλαδή την ανεπάρκεια των εισοδημάτων και τον ακατάλληλο τρόπο με τον οποίο γίνεται η εμπορευματοποίηση των προϊόντων του τομέα. Επίσης ε, προτείνω κάποια μέτρα που έχουν να κάνουν με την διευκρίνηση της ενημέρωσης στους ε, καταναλωτές και για να μην επεκταθώ υπερβολικά. Θα αναφερθώ σε κάποιες, δεν θα αναφερθώ μεμονωμένα σε αυτές τις προτάσεις ε, και θα σταματήσω ε, εδώ. Σας ευχαριστώ. Έχει τον λόγο πρώτος ο Κρίστοφερ Φιέλνερ και κατόπιν ο Μάριο Πέτελο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχω σίγουρα περισσότερες απόψεις από ό,τι είχα για τις δύο προηγούμενες εκθέσεις. Θα προσπαθήσω να ε, περιοριστώ και να σας παρουσιάσω μια γενική θέση καταρχήν. Όσον αφορά την πρόταση αυτή για την ε, κοινή οργάνωση αγοράς ε, του συναδέλφου, πιστεύω ότι είναι πολύ... Βλέπουμε πολύ λίγη αγορά και πολύ δημόσιο χρήμα. λέμε ότι δεν πρέπει να επενδύουμε περισσότερα χρήματα σε κακές υποθέσεις. Εδώ βλέπουμε περισσότερα χρήματα για έναν τομέα που ε, έχει ε, λάβει πολλές ενισχύσεις και μάλλον έχει δημιουργήσει προβλήματα παρά τα έχει λύσει. Η ιδέα ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να διατηρήσουμε την, ε, την, ε, τις κανονικές λειτουργίες της αλληλείας νομίζω ότι είναι λάθος. Η, υπερβολική αλληλευτική ικανότητα στο, στην Ευρώπη έχει να κάνει πολύ με τις ενισχύσεις που έχει λάβει ο τομέας αυτός. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε το βασικό θέμα του εισηγητή είναι να αυξήσουμε τις ενισχύσεις. Ε, αυτό απλά θα ε, επιδεινώσει το πρόβλημα. Αυτά. Τελεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φερέρα για την γνωμοδότησή του που προσφέρει διάφορες ε, ε, διάφορα λαβές για προβληματισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μικρή ε, παράκτια αλία που συχνά είναι οικογενειακού χαρακτήρα. Σε πολλές περιοχές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτού του είδους η αλία, τόσο για, λόγω των απασχολούμενων σε αυτή και όσο και διότι σε πολλές περιοχές είναι η μόνη επαγγελματική διέξοδο Θα πρέπει λοιπόν να αναλυθεί αυτή με το σύνολο του πακέτου μεταρρυθμίσεων για την κοινή αλληλευτική πολιτική που όπως γνωρίζουμε έχει προσανατολιστεί σε μια πιο βιώσιμη αλληλεία ε, που θα προστατεύει το περιβάλλον και θα βοηθά και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Άρα λοιπόν θεωρώ πως οι οργανώσεις των παραγωγών εδώ μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο για να σταθεροποιήσουν τις αγορές και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των ε, παραγωγών, αλλά κυρίως λόγω της συμβολής που μπορούν να κάνουν για τη διαχείριση των απορρίψεων, των ε, αλλιευμάτων, για την επίτευξη του μέγιστου βιώσιμου ε, αποθέματος μέχρι το 2015. Αν και είναι δύσκολο, είναι εφικτό. Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν καλύτερα τα αλλιεύματα σε συγκεκριμένα αποθέματα, ιδιαίτερα αυτά που δεν προορίζονται οπωσδήποτε για εμπορευματοποίηση. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει διεθνή συνεργασία για να μπορούν καλύτερα να ανταγωνιστούν οι εταιρείε, να διαχειριστούν τις ποσοστάσεις και για να γίνει η περιφερειοποίηση που προβλέπεται από τη μεταρρύθμιση. Ο συνάδελφος Φερέρα προτείνει μήνυμο μέτρα αποζημίωσης για να καλυφθεί το κόστος της εκφόρτωσης των ανεπιθύμητων ε, ε, αλλιευμάτων ενώ η Κομισιόν προτείνει δωρεάν ε, ε, ε, παροχή αυτών των παραλιευμάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και αυτές οι δύο λύσεις με βρίσκουν σύμφωνο. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε ένα συνδυασμό των δύο. Πάντως ούτως ή άλλως θα έπρεπε να προβλεφθούν αποζημιώσεις για το κόστος αυτών των παραλιευμάτων και επίσης θα έπρεπε να εμβαθύνουμε περισσότερο στο θέμα που είναι πολύ περίπλοκο όσον αφορά τις ετικέτες, την ετικετοθεσία, όπου θα πρέπει να, φτά, να βοηθούν τον καταναλωτή να προβαίνει σε μια όριμη επιλογή. Ε, αυτό δεν αφορά μόνο το φρεσκάδα του προϊόντος, γιατί αν αυτό αλλιευθεί και διατηρηθεί σε ψήξη ή σε κατάψυξη, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι υγιές για τον καταναλωτή απαραίτητος. Επίσης με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι αυτός ο κανονισμός για την ΚΟΑ που θα έπρεπε να θέσει τις βάσεις για να δώσουμε κάποιες ελάχιστες ενδείξεις για την διεθνή πτυχή της αλληλείας, λείπει εδώ. Κατανοώ ότι η Κομισιόν δεν θέλησε να αντιμετωπίσει αυτή την πτυχή στην πρότασή της, αλλά θεωρώ πως είναι σημαντική αναφορά στην εφαρμογή του κανόνα προέλευσης. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές, από πολλές χώρε εισάγονται προϊόντα της αλίας που δεν υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες ε, που διεθνείς στόλοι ε, αλλιεύουν, δηλαδή και ευρωπαϊκός στόλος ο κανόνας προέλευσης, εάν δεν εφαρμοστεί, θα υπάρχει, αντικυ... θα υπάρχει συνταγωνισμός. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μια ετικέτα που θα ε, καλύπτει αυτήν την ε, έλλειψη και θα υποδεικνύει πού έχει αλλιευθεί το κάθε ε, ψάρι. Να πω και για την Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, που τα χαρακτηριστικά τους είναι διαφορετικά, πολύ διαφορετικά και χρειάζεται να τις αντιμετωπίσουμε επιχωριστά. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση και θα ακούσω ευχαρίστως και τις παρεμβάσεις των άλλων συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα. Τον λόγο έχουν οι πράσινοι. Παρακαλώ. Ο κύριος Άκχαουτ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ λακωνικός γιατί είχαμε εκτενέστατη συζήτηση στην προηγούμενη, συζή... στην γνωμοδότηση αλλά και αυτό το θέμα είναι σημαντικό για την κοινή οργάνωση αγορών. Είναι σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει σαφέστατα στην πρότασή της ότι στόχος της ΚΟΑ είναι να υλοποιήσει τους ευρύτερους στόχους ε, της αλληλευτικής πολιτικής. Είναι σημαντικό να εμείνουμε σε αυτό για να γιατί ε, αρχίζουμε να λέμε ότι πρόκειται η κοινή οργάνωση αγοράς που εξυπηρετεί περισσότερο την αλληλεία παρά την διαφύλαξη των αλληλευτικών πόρων, κάτι που επίσης είναι σημαντικό. Βέβαια, έχουμε κάποιε επικρίσεις προς την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δίνει μεγάλη εξουσία στις οργανώσεις παραγωγών. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε επικριτικοί από το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό, κάτι που κάνει ο εισηγητής και το επικροτούμε, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτό που λείπει από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η σαφής δήλωση ότι θα πρέπει να επιβραβευθούν οι καλύτεροι αλληλείς, αυτοί που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ αυτοί που έχουν κακές επιδόσεις θα πρέπει να, α, έρχονται, να τιμωρούνται κατά κάποιο τρόπο. Σε ό,τι αφορά την εμπορευματοποίηση των παραλιευμάτων. Ε, νομίζω ότι θα, κάνουμε, θα οδηγήσουμε τους ε, σε καλύτερη και επιλεκτικότερη αλία για να μην έχουν απώλειες. Συμφωνώ με τον εισηγητή σε αυτό. Και τέλος μία μικρή προσθήκη ενημέρωση προς τους καταναλωτές. Στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, μιλούμε για τις περιοχές ε, ΦΑΟ. Ε, για να δίνονται περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές ε, από πού προέρχονται τα ψάρια. Βέβαια, η περιοχή αυτή είναι τεράστια ε, και δεν δίνει ουσιαστικά πληροφορίες στους καταναλωτές για το από πού προέρχονται τα ψάρια. Περισσότερες πληροφορίες θα θέλαμε λοιπόν, πιο συγκεκριμένες και συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση. Και τέλος μια ερώτηση στον εισηγητή. Γιατί στην τροπολογία 11α διαγράφει την ευκαιρία να δοθούν κάποια παραλίευματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Γιατί διέγραψε αυτή την πρόταση από την τροπολογία του ο εισηγητής. Τελευταία ομιλήτρια, Ιαννα Ρόσπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Χαίρομαι που ο εισηγητής σκέφτεται τη βιωσιμότητα και την ε, οικολογία και την ε, υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα με την προσοχή που δίνει στην υδατοκαλλιέργεια, διότι ε, αυτός ο τομέας θα μπορέσει να ελαφρύνει την πίεση στην παράκτια αλληλεία. Ο εισηγητής μιλάει για βιωσιμότητα, δηλαδή να αποφύγουμε την υπεραλίευση. Αλλά όλων τούτων λεχθέντων Έχω και διάφορες αναμνήσεις όσον αφορά την, ε, την ε, χρηματοδότηση. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για μένα. Ε, η αλληλεία και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας είναι για μένα ένας τομέας οικονομικός και θα πρέπει να σταματήσουμε όλες αυτές τις επιδοτήσεις. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο Φιέλνερ η ομάδα ECR θα κοιτάξει πιο προσεκτικά την ε, έκθεση αυτή, να δούμε αν μπορέσουμε να βρούμε κοινό τόπο, αλλά γενικά πιστεύω ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα εξέβρεσης των οικονομικών πόρων για να στηρίξουμε έναν κανονικό εμπορικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Άννα Ρόσπαχ. Να δώσω τώρα την δυνατότητα στην Κομισιόν να απαντήσει στη συζήτηση από τη Γενική Διεύθυνση. Μάρε, έχουμε τον κύριο Ράμπερτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα τρία σημεία που είναι διευκρινιστικά. Καταρχήν, Μιλούμε για ένα στοιχείο που, απαιτεί, που αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα, τμήμα της αναθεώρησης της κοινής πολιτική. πολιτικής. Ευθυγραμμίζεται δηλαδή πλήρω με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε και ε, εντό ολίγου θα ασχοληθείτε και με τη χρηματοοικονομική δημοσιονομική πτυχή, όπω είπατε και προηγουμένω. Πρόκειται λοιπόν για ένα αναπόσπαστο στοιχείο, για μια ψηφίδα του πάζλ, αυτού του ψηφιδωτού. Και η κόα των αλευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργεια έχει δύο άξονες. Καταρχήν επιτρέπει την οργάνωση των κλάδων αλίας και υδατοκαλλιέργειας, ηχθειοκαλλιέργειας και δεύτερον ε, μιλά για την εμπορευματοποίηση των ε, προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας, ηχθειοκαλλιέργειας. Ό,τι αφορά ε, τον πρώτο στόχο, τον πρώτο άξονα, στόχος είναι να δώσουμε στον κλάδο την ευκαιρία να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει πραγματικά υπεύθυνο ε, παράγων στην εξασφάλιση βιώσιμη αλληλεία. Γιατί πραγματικά αυτοί είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται καθημερινά με το ζήτημα αυτό και εφαρμόζουν εμπράκτο την αλληλευτική πολιτική που θα αποφασίσουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, θα συναποφασίσουν μάλλον. Τι προτείνουμε λοιπόν στην αναθεώρηση τη ΚΟΑ. Προτείνουμε μια ρηξικέλευθη αναθεώρηση ε, τον τρόπο οργάνωσης αυτών των παραγωγών. Γιατί πριν από 40 χρόνια στόχος αυτών των οργανώσεων ήταν να, διαχειριστούν τις παρεμβάσεις στην αγορά. Τώρα πια προτείνουμε αυτές οι οργανώσεις παραγωγών να συμμετέχουν και ενεργά στην προαγωγή μιας αηφόρου αλίας. Και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για να ελοπιθεί αυτός ο στόχος, επαναλαμβάνω, προτείνει κάποια μέσα, όχι μόνο δημοσιονομικά, και ουσιαστικά δίνει μια εργαλειοθήκη στις εργανώσεις παραγωγών για να διαχειριστούν καλύτερα και να υλοποιήσουν αυτό το στόχο της αηφόρου αλίας. Ένα άλλο στοιχείο που είναι και το πιο καινοτόμο της πρότασης είναι ότι σε αυτή την εργαλειοθήκη που δίνουμε στου οργανώσει παραγωγών επιμένουμε στην ε, σύσταση ενός νέου συστήματος που φέρνει τις οργανώσει παραγωγών στο επίκεντρο και του δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τις, ε, την παραγωγή των μελών του και να διευκολύνει τη διάθεση των προϊόντων του. Αυτό ισχύει και για την αλία και για την ε, είδα το για να μπορέσουν οι αελείς να ψαρεύουν και οι ε, να εκτρέφουν ε, ψάρια. Και μάλιστα το σύστημα αυτό είναι εθελοντικό. Τα μέλη δίνανται να συμμετέχουν σε αυτό την οργάνωση που θα οργανώνει καλύτερα τις δραστηριότητες των μελών της. Αυτά εν είδη προημίου. Τώρα θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ε, επιμέρους ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο για την ε, βιοτεχνική Ελία. Την Ελία μικρής κλίμακος. Η πρόταση της ΚΟΑ συνάδει πλήρως με το στόχο προάσπισης ε, της ε, αλίας μικρής κλίμακος και οι οργανώσεις παραγωγών είναι κατεξοχήν οι οργανώσεις συλλογικής διαχείρισης αυτών των μικροαλιαίων και είναι και το πιο αποτελεσματικό επίπεδο διαχείρισης. Και μάλιστα στις πληροφορίες στους καταναλωτές προσθέσαμε και την ημερομηνία αλίευσης. Βέβαια κάποιος εξέφρασε αντιρρήσει για αυτό το στοιχείο. Επαναλαμβάνω, είναι ένα καινοτόμο στοιχείο της ενημέρωσης ε, του καταναλωτή για προϊόντα αλίας και δατοκαλλιέργεια. Στόχος μας είναι να γίνει μια διαφοροποίηση των προϊόντων που αλλιεύθηκαν πριν από τρει μέρες από αυτά που αλλιεύθηκαν πριν από τρει εβδομάδες. Δέχομαι πλήρω τι παρατηρήσει. Ε, τον προλαλισσάντων που είπαν ότι το, ε, το γεγονός ότι ένα ψάρι είναι φρέσκο δεν σημαίνει ότι είναι και πολύ κέρι του ποιότητα. Αλλά αυτό θα το δει ο καταναλωτή που θα διαλείπει. Η κεφάλαια είναι ε, σε κακή κατάσταση, αλλά θα ξέρει πότε αλλιεύτηκε. Και νομίζω ότι έτσι ευνοούμε την αλληλεία εγκύτητα ε, από την αλία που είναι βιομηχανική ή βιομηχανική και που είναι πολύ πιο μακριά από τον καταναλωτή. Έτσι εξασφαλίσουμε και συνθήκες ε, ίσου ανταγωνισμού σε σχέση και με τα εισαγόμενα προϊόντα. Ε, αναφέρθηκε η διάλυση των μηχανισμών και των εργαλείων. Εδώ δεν μιλούμε μόνο για νέες επιδοτήσεις. Σε ό,τι αφορά την κοινή οργάνωση αγορών, έχουμε δύο δημοσιονομικά μέσα. Έχουμε και το ενιαίο δημοσιονομικό μέσο, αλλά έχουμε και δύο άξονες. Ο πρώτος είναι οι παρεμβάσεις με την αμυγένεια και εκεί προτείνουμε μια σταδιακή κατάργηση, phasing out. Όχι λοιπόν δεν θα δοθούν πια χρήματα για καταστροφή ψαριών, κάτι που γίνεται εδώ και 40 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα οι παρεμβάσει που θα επιτρέπονται για, ως ενίσχυση για την αποθεματοποίηση θα επιτρέπουν όχι μόνο να αποφεύγει την καταστροφή του ψαριού, αλλά να ε, του δίνουμε και μια προστιθέμενη αξία. Λογική μας λοιπόν είναι ο προσανατολισμός μας προς την αγορά για την αναθεώρηση αυτή. Και λέμε 45 εκατομμύρια ευρώ για, για μία πενταετία, μέχρι ότου ε, ολοκληρωθεί η μελέτη των επιπτώσεων, ώστε τα περίφημα σχέδια παραγωγής και θέσης εμπορία να αποφέρουν τους καρπούς τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά Α, το θέμα ε, της, ε, του διαχωρισμού σε ζώνες και την ένδειξη της ζώνης ο καταναλωτής σήμερα δεν είναι και πολύ ενημερωμένος όταν μια ετικέτα αναφέρει βορειοανατολικός Ανατολικό-τελετικό. Ξέρω αν γνωρίζει τι σημαίνει κάτι τέτοιο ο καταναλωτής. Δεν είναι ότι ε, αναφέρεται ζώνη ΦΑΟ, δηλαδή ζώνη 12. Στο μέλλον προτείνουμε να αναφέρονται όχι μόνο ζώνες, αλλά και ε, διαιρέσεις ή υποδιαιρέσεις. Δηλαδή, μπορεί να αναφέρεται ότι το ψάρι είχε αλλιευθεί στη Βόρεια Θάλασσα, στην θάλασσα της Ιρλανδίας, στο Βυσκαϊκό κόλπο και ούτω καθεξής. Και καλύτερα αυτό να το κάνουμε με ετικέτες παρά με κώδικο. Σε ό,τι αφορά την προαγωγή για την αλλιεύση νεαρών ψαριών ηχθιδίων. Λάθος. Στην αποστολή που αναθέτουμε στις οργανώσεις παραγωγών, προβλέπετε ότι μπορούν ταυτόχρονα να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα προκειμένου να μειωθεί και σταδιακά να καταργηθεί, να εξαλειφθεί τελείως η αλίευση ηχθιδίων. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Όπως είπα όμως, θέλουμε και μια συνέπεια και συνοχή. Εν αναμονή της ολοσχερούς κατάργησης ε, των απορρίψεων θα θέλαμε η οργανώσεις παραγωγών να εξασφαλίσουν την σωστή εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται και στο Συμβούλιο για την διάθεση των απορρίψεων. Δεν υπάρχει καμία αμφισημία. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δώσουμε ναύσματα για την αλίευση νεαρών ψαριών, ηχθιδίων ή αντίστοιχων προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την διανομή σε φιλαθροπικούς ε, οργανισμούς ή για αγαθοργούς σκοπούς, ίσως η έννοια της φιλαθροπίας ε, δεν είναι ε, κάτι για το οποίο υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Τι θα πει φιλαθροπικό σκοπός ή φιλαθροπικό ίδρυμα. Ίσως αυτό το σημείο χρήζει ε, για να δούμε τι εννοούμε με τέτοια δωρεάν διανομή σε φιλαθροπικά ιδρύματα. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία ως προς την φρεσκάδα του ψαριού τα ανέφερα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχω απαντήσει πια. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Για το διακρατικό χαρακτήρα. Ένα από τα πράγματα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακριβώς η ανάπτυξη αυτού του στοιχείου, γιατί η διακρατικότητα ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να φέρουμε τους φορείς ε, στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Στο παρελθόν είχαμε κάποια παραδείγματα και αιτήματα που τελικά δεν ευωδόθηκαν. Ακριβώς επειδή το κοινοτικό πλαίσιο δεν διευκόλυνε την εφαρμογή μιας τέτοιας διακρατικής δυναμικής. Πολλά δε μάλλον που τα ψάρια έχουν αυτή την ενοχλητική τάση να μην ε, αναγνωρίζουν σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ε, θέλει να, να προωθήσει κάτι τέτοιο και σε διακλαδικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανώσεων παραγωγών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ο εισηγητής θέλει να πάρει πάλι το λόγο. Παρακαλώ. Μάλιστα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι συνοπτικός. το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί στην Επιτροπή Ελίας, μετά που θα κάνω τα σχόλιά μου θα μεταβώ εκεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους που θα ληφθούν ε, δεόντως υπόψη. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών, ότι είμαι στη διάθεσή σας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για τις τροπολογίες ε, ε, για να εξετάσουμε διεξοδικά και εμβριθέστατα με κάθε σκιώδη συγητή οποιασδήποτε τροπολογίες. Τώρα, ω προ τα σχόλιά σα, ο κύριος Φέλντερ του ΕΛ και η κυρία Ρόσμπαχ μίλησαν για το γεγονός ότι ίσως με την πρόταση αυτή αυξηθούν οι επιδοτήσεις και τα κρατικά κονδύλια που αφιερώνονται στην Αλία. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι έχω μία ε, ανισχύει και την πρόταση αυτή. Η μέλημά μας είναι να ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε το εισόδημα των αλλαίων. Γιατί πιστεύω ότι αν ε, αναβαθμιστεί, αν αναγνωριστεί η ελευτική προσπάθεια και αν ε, αμείβονται δίκαιοι για, την, για τον κόπο τους οι αλλοίς, νομίζω ότι θα αλλιεύουν και λιγότερο σε τελική ανάλυση. Πάντως, Υπάρχουν πολλές και διάφορες προτάσεις για την υλοποίηση του στόχου της βελτίωσης του εισοδήματος των αλλιών και δεν είναι όλες αυτές οι προτάσεις που προϋποθέτουν αύξηση των κρατικών κονδύλιων. Υπάρχει μια πρόταση που προβλέπει και το μόνο που κάνει είναι να ε, επιδιώξει μια πιο ακριβωδίκη κατανομή της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα. Γιατί αυτή τη στιγμή η κατανομή είναι άνηση και άδικη ε, στους διάφορους κρίκους έλιας, στους διάφορους κρίκους οι περισσότεροι τα περισσότερα κέρδη τα καρπώνονται οι μεσάζοντες προτείνουμε λοιπόν ένα μηχανισμό επέμβαση σε αυτή την αλυσίδα για να εξασφαλίσουμε πιο ακριβωδική κατανομή των εισοδημάτων σε όλους τους κρίκους της αλυσίδα. κάτι τέτοιο δεν προϋποθέτει αύξηση των κρατικών κονδύλιων ή των επιδοτήσεων απλώς μια δικαιότερη ένα δικαιότερο καταμερισμό. Υπάρχουν και οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Και ας μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι θετικοί εξωτερικοί παράγοντες και περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί που σήμερα δεν επιβραβεύονται δεόντως ή δεν αμείβονται δεόντως, δεν αμείβονται δεόντως από την αγορά. Γι' αυτό και χρειάζονται επιδοτήσεις. Εκτός και αν θέλουμε να θυσιάσουμε αυτούς τους θετικούς εξωτερικούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες, αλλά και μια τέτοια επιλογή θα έχει κόστος. Εγώ θεωρώ ότι η περιβαλλοντική στόχη και ιδιαίτερα ο στόχος ε, του, της κατάργησης των απορρίψεων είναι πολύ σημαντικός και αξιέπαινος. Θέλουμε ένα μηχανισμό που θα εξασφαλίζει την ευκολότερη υλοποίηση του στόχου, αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο να ολοποιήσουμε του στόχου. Και συμφωνώ με τον κύριο Πυρίγιο ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να προέλθει από, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελίας και Θάλασσα και ναυτιλιακών θεμάτων. Αλλά θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα και τη ΣΚΟΑ να χρηματοδοτεί τέτοιου είδου μέτρα. Παρόλο μπορεί, που μπορεί κάποια κονδύλια να προέλθουν και από άλλο χρηματοδοτικό μηχανισμό. Έστω και ελάχιστα θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την κατάσταση. Να ε, στηρίξουμε τον κόστο δηλαδή ε, για την αποθεματοποίηση αυτών των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων. Έστω και ελάχιστα θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτή την αποθεματοποίηση, όσο το απαγορευθούν οι απορρίψεις. Γιατί επαναλαμβάνω, άλλο η θέσπιση στα χαρτιά και άλλο η έμπρακτη εφαρμογή. Εμείς θέλουμε και μηχανισμούς που θα εξασφαλίζουν έμπρακτη εφαρμογή αυτών που θεσπίζουμε στα χαρτιά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Ο Μπάτς Έκχαουτ ε, με ρώτησε γιατί διέγραψε τη δωρεάν διανομή εκφορτωθέντων προϊόντων σε φιλαθροπικά ιδρύματα για καθοεργούς σκοπούς. Δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Και επειδή διαγράφεται από εδώ δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Απλώς ε, επειδή κάποιες οργανώσει παραγωγών εξέφρασαν ανησυχίε, δεν θα ήθελα να αναφέρεται κάτι τέτοιο ω υποχρέωση, υποχρέωση δηλαδή των οργανώσεων παραγωγών να κάνουν δωρεάν διανομή. Γιατί εξαιτία των χαρακτηριστικών και του μεγέθου του, δεν έχουν τη δυνατότητα για δωρεάν κατανομή όλε οι οργανώσει των ε, παραγωγών. Αυτά κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι κάλυψε τα περισσότερα στοιχεία. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε ε, να θυσιάσουμε όλες τις παρεμβάσεις στην αγορά, ακόμη και όταν είναι μικρής εμβέλειας και έξυπνες. Γιατί έτσι μπορεί να θυσιάσουμε την παράκτη, τη βιοτεχνική αλληλεία και να αμελούμε συγκεκριμένες διαστάσεις περιβαλλοντικές και κοινωνικές που μας εξυπηρετούν και που δεν ανταμείβονται δεόντως από την αγορά. Δεν θέλουμε να χάσουμε αυτούς του εξωτερικούς παράγοντες. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος που ακολουθεί μερικέ φορέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. Ολοκληρώσαμε έτσι τη συζήτηση ε, της έκθεσης αυτής ε, στην ΕΝΒΗ. Θα ψηφίσουμε 25-26 Απριλίου, 9 ε, Μαρτίου, 12 ε, η ώρα είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. και στην Επιτροπή Αλίας που είναι αρμόδια επί της ουσίας ε, θα γίνει ψηφοφορία στις 30 ε, Μαΐου και στην Ολομέλεια 2 με 5 Ιουλίου. Ε, σημαντικό το θέμα, ιδιαίτερα για τους ε, συναδέρφους ε, που έχουν αλληλεία στην εκλογική τους περιφέρεια, διότι εκεί θεωρείται η αλία όχι μόνο επαγγελματικό κλάδος, αλλά είναι και μέρος της πολιτιστικής παράδοσης. Όλα αυτά λοιπόν συνοψίζονται στο πακέτο περί και Έχουμε γι' αυτό και την ευθύνη να ε, πετύχουμε στο θέμα αυτό, διότι είναι θέμα πρακτικής πολιτικής. Φτάνουμε έτσι στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι το 7 τροποποίηση της, ε, του κανονισμού 1185 του 2003 σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους. Η συγητής είναι ο συνάδελφος Αντρέας Ανώνη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλήσαμε για πολλά προβλήματα της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο είδος και τα προβλήματά του, τους καρχαρίες. Από το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση εθέσπισε ένα κανονισμό για να απαγορεύσει την πρακτική της ε, αφαίρεσης των πτερυγίων επί του σκάφους ε, και της ρήψης του σώματος στην θάλασσα. Όμως αυτός ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης εξαιρέσεων για ειδικέ άδειε, ε, εξαιρέσεις που, αφορούν, που επιτρέπουν μάλλον εκεί την αφαίρεση πτερυγίων επί του σκάφους. Συγκεκριμένα αυτές οι ειδικέ άδειε θα έπρεπε να είναι εξαιρέσεις, ωστόσο αποτέλεσαν τον κανόνα, ιδίω για δύο κράτη-μέλη, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακόμα και αν ε, πρόκειται για μία μόνο ε, έγκριση. Αυτό το σύστημα της έγκρισης των εξαιρέσεων δημιουργεί επιπλοκές γιατί αφορά το όριο της αναλογίας 5% για την αφαίρεση των πτερυγίων επί του σκάφους. Είναι ένας κανόνας που πολύ δύσκολα μπορεί να εξακριβωθεί ε, και να ελεγχθεί. Γιατί εξαρτάται από το αν έχουν αφαιρεθεί τα σπλάχνα, αν έχει αφαιρεθεί το κεφάλι ή το δέρμα και επίσης ε, μπορεί το βάρος του σώματος να ε, διαφέρει ανάλογα με το είδος του καρχαρία. Άρα λοιπόν μπροστά σε όλα αυτά τα προβλήματα συμφωνήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο και απαραίτητο να εισαχθεί υποχρέωση εκφόρτωσης των καρχαριών ε, με τα πτερίγια φυσικά συνδεδεμένα με το σώμα. Μετά από αυτή την επιστημονική διαπίστωση και μετά από τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον ΦΑΟ, η Κομισιόν το 2009 παρουσίασε το κοινό σχέδιο δράσης για τη διατήρηση και τη διαχείριση των ε, καρχαριών, όρια της οποίας είναι και αυτή η πρόταση που προβλέπει την κατάργηση όλων των εξαιρέσεων που προβλέπονται σήμερα, των ειδικών αδειών δηλαδή. Ε, για να διευκολυνθούν οι αλληλείς προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κοπής των πτεριγίών με τρόπο ώστε να είναι ακόμα ε, προσκολλημένα στο σώμα ώστε να διευκολυνθεί η αποθήκευση. τα ψάρια που ανήκουν στην ταξινομική βαθμίδα των ελασμοβραχίων που περιλαμβάνονται οι καρχαρίες και τα σελάχια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα βιολογικά όντα τα, γιατί έχουν πολύ χαμηλό ρυθμό αναπαραγωγής. Να φανταστείτε ότι ένα από αυτά τα είδη, το, η μάκο, οι καρχαρίε μάκο, φτάνουν στη σεξουαλική οριμότητά του στα 7 με 9 έτη, ενώ το θηλυκό φτάνει σε τέτοια οριμότητα στην ηλικία των 19 με 21 ετών. Πέρα από τα αστεία που έλεγε πριν ο συνάδελφος Ντέιβις, αυτά τα είδη κινδυνεύουν να μην φτάσουν ποτέ σε ηλικία σεξουαλικής οριμότητας. Ε, επιπλέον αναπαράγονται μόνο κάθε τρία χρόνια και έχουν περίοδο κύησης 15 με 18 μήνες για, ε, γεννούν πολύ περιορισμένο αριθμό μικρών. Όσον αφορά τα είδη που αλλιεύονται περισσότερο είναι ακριβώς σε επίπεδο ε, στην Ισπανία έχουμε το 50% των γλαυκοκαρχαριών που αποτελούν που το καρχαρία που είναι και γνωστός ως ε, μπλε καρχαρίας και το 10% καλύπτεται από το είδος μάκο. Μιλάμε για 78% γλαυκοκαρχαρίες. Τώρα, η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης, η IUCN, θεωρεί τον καρχαρία μάκο το είδος και το γλαύκο καρχαρία ως σχεδόν απειλούμενο στον κόσμο και ευάλωτο στη Μεσόγειο. Εν ώψη λοιπόν της μείωσης αποθεμάτων των ειδών αυτών, πολλές χώρες έχουν αυτόνομα αποφασίσει να μην επιτρέπουν πλέον την αφαίρεση πτερυγίων επί των σκαφών. Όπως ε, χώρες αυτές είναι η ΙΠΑ, η Ταϊβάν, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι έχουν συμβάλει στο να αποφευθεί όντως να η κοπή, η αφαίρεση των πτερυγίων επί των σκαφών και η ρήψη των σωμάτων στη θάλασσα. Το 2009 μιλάμε για 111.000 τόνους καρχαριών και σελαχιών που έχουν εκφορταθεί σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΦΑΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από του μεγαλύτερου εξαγωγεί περιτυχίων ε, καρχαρία προ αγορέ του Χονγκ Κόνγκ και τη ε, Κίνα. Και αυτό το εμπόριο είναι πολύ επικερδές γιατί τα πτερίγια είναι το βασικό συστατικό τη περιζήτητη κινέζικη σούπα που πωλείται στη συνέχεια σε πολύ ψηλέ τιμέ. Πράγμα το οποίο φυσικά δίνει κίνητρα για αυτό το είδο στην Τώρα, όσον αφορά την, έκθεση της, την πρόταση μάλλον της Επιτροπής, θεωρούμε πως είναι σωστή. Εγώ έχω εισάγει μόνο κάποιες τροπολογίες για να διευκρινίσω κάποια στοιχεία, κάποια τμήματα και για να ενισχύσω αυτή την απόλυτη απαγόρευση χωρίς εξαιρέσεις για την αφαίρεση των πτερυγίων ε, πάνω στα σκάφη. Πιστεύω πως είναι δίκαιο να βάλουμε επίσης, να προβλέψουμε οι εξαιρέσεις να γίνονται, μάλλον η αφαίρεση να μην γίνει μόνο, μάλλον η απαγόρευση αυτή να μην ισχύσει μόνο για τα ευρωπαϊκά ελευτικά σκάφη, αλλά και για όλα τα άλλα σκάφη που εκφορτώνουν στα λιμάνια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί υπάρχουν περιπτώσει ε, όπω στο Βίγκο ή στη Γαλλική ή στο Λασπάλμα, όπου φτάνουν τα ιαπωνικά παραγαδιάρικα και ξεφορτώνουν εκεί. Έχουμε επίση λάβει υπόψη τεράστια έλλειψη επιστημονικών δεδομένων για τα ίδια αυτά. Και άρα πιστεύω πω ήταν δίκαιο να μην περιοριστούμε στην παρακολούθηση των ποσοτήτων και το βάρος των αλλιευμάτων, αλλά τα είδη και τα είδη ε, που αλλιεύονται, το, καθώς και ε, το συνολικό βάρος και για κάθε περιοχή αλλιώς, ώστε να δημιουργηθούν επιστημονικώς ορθές βάσεις δεδομένων που είναι αναγκαίε για την εφαρμογή των μέτρων που θα αποσκοπούν στην ελληνοποίηση του κοινοτικού σχεδίου δράση για τη διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση των καρχαρίων. Επίση, θα πρέπει να παρακολουθούμε την ποιότητα των ελέγχων που γίνονται, ε, γιατί έτσι ώστε να έχουμε πληροφορίε σχετικά με τι επιθεωρήσεις και τι κυρώσει που εφαρμόζονται στα διάφορα κρατή-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποιο ελεγκτικό σώμα και τέτοιες περιπτώσει, όπω αυτή που αναφέρθηκε ο ο, ο Chris όπου αλλιεύθηκαν ε, αλλιεύματα ε, αξίας 60 εκατομμυρίων λιρών στερλίνων είναι μάλλον μόνο η κορυφή ενός παγόβουνου και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε την προβληματική των παραβιάσεων, των ελέγχων και των κυρώσεων. Θέλησα επίσης να βάλω στο διατακτικό τον ορισμό του γεγονός ότι θα πρέπει ε, τα πτερίγια να βρίσκονται σε φυσική συνοχή με το σώμα, γιατί στο κείμενο μέχρι σήμερα απλώς αυτό υπονοείτο, και επίσης να βάλουμε τη σημαντική πολιτική στήριξη που υπάρχει για πλήρη απαγόρευση της αφαίρεσης των πτερυγίων στο, των καρχαριών εδώ στο Κοινοβούλιο. Γιατί το 2010, στις 16 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκε γραπτή δήλωση από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών που, προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση της αφαίρεσης των πτερυγίων των καρχαριών ε, πάνω στα σκάφη. Πιστεύω λοιπόν πως είναι μια πρόταση πολύ σημαντική που θα πρέπει να τη στηρίξουμε και αν και πιστεύω πως είναι ένα ακόμα βήμα προς την προστασία και το τέλος της ε, εξαγωγής των ε, της αφαίρεσης μάλλον των πτερυγίων, ακριβώς επειδή το αδύναμο σημείο είναι η έλεγχη. Σίγουρα αυτό θα ε, θα βοηθήσει τις θάλασσες, τους καρχαρίες αλλά και τους αλείς, γιατί αυτό σημαίνει προστασία των αποθεμάτων αυτού του είδους των ε, ψαριών. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Τζανόνη. Να κάνω την εξή πρόταση. Οι σκιώδεις ε, να πάρουν το λόγο για 2,5 λεπτό και οι υπόλοιποι για 1,5 λεπτό, διότι αλλιώς δεν θα προλάβουμε καθόλου και έχουμε και άλλο ένα σημαντικό θέμα στην ημερησία διάταξη όπου έχουμε προσκαλέσει την Κομισιόν. Ε, θα ήθελα λοιπόν να τηρήσουμε το χρόνο. Εάν ε, συμφωνείτε θα προχωρήσουμε έτσι. Ε, λοιπόν, ε, η πρώτη ομιλήτρια έχει 2,5 λεπτά το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήμουνα, ε, συνυπέγραψα την δήλωση ε, του 2010 για την αποκοπή των πτεργείων των καρχαριών και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που έχουμε τώρα αυτή την πρόταση από την Κομισιόν. Πρόκειται για μια πρόταση η οποία στόχο έχει να καλύψει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τις οποίες υποδείξαμε με την διακήρυξή μας για τον κανονισμό για την αποκοπή των πτερυγίων ε, των, καρχαριών. Αυτό είναι σημαντικό θέμα για την βιοπικιλότητα ε, και για τα οικοσυστήματα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καρχαρίες με την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολύ ισχυρό μέσο. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που έχουμε τώρα αυτή την έκθεση διότι ενισχύει την προηγούμενη πρόταση της Κομισιόν και θα ήθελα να προτείνω να αντιψηφίσουμε τις ε, τροπολογίες που αποδυναμώνουν την πρόταση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους κανόνες αυτούς και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ε, διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ε, με αυτήν την διατήρηση θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και την βιώσιμη αλληλεία. Στηρίζω λοιπόν την πρόταση και επαναλαμβάνω ότι συνυπέγραψα και συν, ε, ε, συνέγραψα επίσης την ε, διακήρυξη που υπέγραψα η οποία υπέδειξε τις ελλείψεις στο σύστημα οι οποίες αποτελούσαν αντικείμενο αρνητικής εκμετάλλευσης. Εκφράζω λοιπόν τη χαρά μου που έχουμε τώρα πια αυτή την πρόταση και ελπίζουμε με την υπερψήφιση να έχουμε μια ακόμα πιο ισχυρή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Η πράσινη τώρα. Η συνάδελφος Μπελιέ, παρακαλώ, δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα έπρεπε να μείνω κάτω από τα δυόμιση λεπτά, γιατί θέλω καταρχήν να συμφωνήσω με την πληρέστατη πρόταση του εισηγητή Τζανόνι και να τον ευχαριστήσω για αυτή την εργασία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ωστόσο των συναδέλφων σε αυτήν την απέσια, την βίαιη και σοκαριστική πρακτική που γίνεται σε ένα είδος τον καρχαρία που βεβαίως ε, χαίρει πολύ λιγότερη στοργής και ενδιαφέροντος από ό,τι διάφορα άλλα θηλαστικά είδη Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι αυτές οι πρακτικές αφαίρεσης των πτερυγίων των, του Καρχαρία, όπως γίνονται από ευρωπαϊκά σκάφη, ε, είναι συγκρίσιμη με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για ε, το εμπόριο ελεφαντοστού που επίση είναι μια φρικτή πρακτική. Επίσης με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι παρά την απαγόρευση αυτή τη πρακτική, οι εξαιρεσει έχουν οδηγήσει 15% ε, ε, των εξαγωγών προς ε, τις καταναλώτερες χώρες είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό καλλιεύματα. Είμαστε στη δεύτερη θέση όσον αφορά την αλίευση καρχαριών και όπως ε, τόνισαν και οι προηγούμενοι, ε, ομιλήτρια θα πρέπει αυτή η πρακτική να σταματήσει. Κάναμε σχετική δήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2010 και στο όνομα των Ευρωπαίων Οικολόγων υποστηρίζουμε απόλυτα τις προτάσεις που γίνονται σε αυτή την πρόταση για να καλέσουμε την Επιτροπή Αλληλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσουν την απόλυτη απαγόρευση αυτών των πρακτικών και την ενίσχυση των ελέγχων έτσι ώστε η βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σταματήσει αυτή η πρακτική να εφαρμοστεί πραγματικά και να πάψει αυτή η σφαγή που θα έπρεπε να μας σοκάρει τουλάχιστον τόσο όσο και η κατάσταση στο Καμερούν με τους ελέφαντες. Σα ευχαριστώ. Και ο Μάρτιν Κέλλναν, ε, αντί για συνάδελφο ε, Ζουλή Καφή για μισή λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, ε, Ματίας, και πάλι. ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της Τζούλη Κέλλιν, θα πάρω το λόγο εκ μέρους της. Να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για τις προτάσεις του. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε την που διαβάσαμε την έκθεση. Ε, προφανώς ο εισηγητής ε, ε, επικροτεί την πρόταση της ε, Κομισιόν, την ενίσχυση της πρότασης της Κομισιόν με την κατάργηση των, των παρεκκλήσεων που υπήρχαν, ε, όπως έχουν πει οι συνάδελφοι, είναι μια πρακτική η οποία υπονομεύει την βιωσιμότητα των, ε, ε της αλληλείας και των ε, οικοσυστήματων. Ε, η ανάκληση των σχετικών αδειών δεν θα εμποδίσουν την εφόρτωση των καρχάριων από τα ε, κράτη-μέλη. Ε, θα πρέπει, ε, όμως, όπως αναφέρει ο εισηγητής στις τροπολογίες του 5, 10 και 15, θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη η επιβολή του νόμου. Όπως έχουν δείξει παρόμοιες παρόμοιοι περιορισμοί σε άλλα κράτη όπως είναι ε, η ΙΠΑ, η Αυστραλία και ε, το η Ταϊβάν. Ε, οποιαδήποτε τέτοιο μέτρο δεν θα είναι εις βάρος του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης ο λόγος ε, πτερυγίων και ε, σωμάτων όπου περιορίζεται το βάρος ε, των πτερυγίων στο 5% του συνολικού βάρους καρχαριών είναι ένα μέτρο το οποίο είναι δύσκολο να επιβληθεί. Είναι ήδη πολύ επίκης ο αυτός όπως αυτό που εφαρμόζεται από άλλους εισαγωγείς. Μία πιθανή λύση όπως αναφέρει η μελέτη επιπτώσεων της Κομισιόν θα ήταν η μεταφορά ε, σε έναν λόγο 5% ε, αλλά σε σχέση με το βάρος ε, των νεκρών ζώων. Το να είναι συνδεμένα με το σώμα του καρχαρία τα πτερίγια μπορεί να αποτελέσει μπορεί να είναι επικίνδυνο για κάποιες περιπτώσεις. Κάποια ψάρια όπως ο Σολομός και ο Ερυθρός Τόνος ε, ε, κόβονται και καταψύχονται ε, στην θάλασσα. Στη θάλασσα πιθανή λύση για το θέμα αυτό είναι η μερική αποκοπή του πτερυγίου και το να διπλώνεται πάνω στο σώμα του καρχαρία. Ευχαριστώ πολύ. Από 1,5 λεπτό ο Κρις Ντέιβις και κατόπιν ο Καρλ Σλίτερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ να περιοριστεί το shark Το είχαμε πει και πριν πολλά χρόνια. Χαίρομαι που επιτέλους, έστω και καθυστερημένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε προς το μέρος μας και συμφωνώ και με τις προτάσεις του κ. Ζανώνη. Σήμερα, με την παρούσα κατάσταση, μπορεί κανείς να ε, εκφορτώσει το σφάγιο, το σώμα του καρχαρία και τα πτερία, αλλά ξεχωριστά. Βέβαια δεν γίνεται σωστή καταγραφή. Και ιδιαίτερα ο γλαφοκαρχαρίας ε, είναι απειλούμενο είδος εξαιτίας της υπεραλίευσης που γίνεται. Βέβαια αμφισβητούνται αυτοί οι δύο ισχυρισμοί από τους πολέμιους του κανονισμού. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν ε, ε, στοιχεία για κακή πρακτική ή για έλλειψη δήλωσης καταχώρησης ούτε και αυτό αποδεικνύεται, και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα αποθέματα γλαυκοκαχαρία. Πολύ αφιβάλλω και για τους δύο ισχυρισμούς για το να ευσταθούν. Τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο εδώ. Είναι δύσκολο να διαχωριστεί το πτερίγιο από το σώμα του καρχαρία, από τη στιγμή που είναι, γίνεται βαθιά κατάψυξη, γιατί είναι στερεό. Εκτός αν μπουν σε ξεχωριστά α, σημεία ή αν αυτό που ζητάμε είναι τελικά να διπλώσουμε το, το πτερίγιο πριν τη βαθιά κατάψυξη ώστε να μπορεί να γίνει ο διοχαρισμός. Σε τέτοια περίπτωση δεν διαφωνούμε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρόταση και χαίρομαι για την διεύρυνση του ορισμού για το TST ε, σκάφος με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα όπως μας ε, περιέγραψε και ο Κρίς Ντέιβις. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με την πρακτική αυτή το να σκοτώνουμε ένα ε, είδος που ούτως ή άλλως αναπτύσσεται πολύ αργά, αναπαράγεται πολύ δύσκολα, και απλώς για να χρησιμοποιήσουμε ένα κλάσμα ουσιαστικά του σώματός του που θεωρείται ως χρήσιμο προϊόν. Πραγματικά αυτή η, πρακτική, το φίνινγκ, είναι απεχθής. Τώρα δεν ξέρω αν έτσι μπορούμε να κόψουμε το πτερίγιο, να το λυγίσουμε, αλλά δεν ξέρω αν κανένα νομομαθή έχει βρει κανένα παραθυράκι στη διατύπωση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν ε, όντω υπάρχει, να το διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Καρλ Σλίτερ. Συγκεκριμένη ερώτηση προ την ε, Κομισιόν. Να τη δώσω ε, το λόγο για τρία λεπτά από την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ, ο Χρήστο Θεοφίλου. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μια ναι, και έχω μόνο τρία λεπτά, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο λακωνικός γίνεται. Είχα πολλά να πω, αλλά χάρη στους προλαλήσαντες καλύφθηκε ένα μεγάλο τμήμα των δικών μου παρατηρήσεων. Θα ήθελα πρώτα να κάνω μια βασική διάκριση μεταξύ της αφαίρεσης του πτερυγίου και της μεταποίησης. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς για το τι έχουμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Το φίνινγκ, η πρακτική αυτή, ε, είναι η αφαίρεση του απτεριγίου και η απόρριψη του σώματος. Από τη στιγμή που αφαιρεί κανεί το πτερίγιο αλλά κρατά το σώμα, αυτό, σημαίνει, αυτό είναι μεταποίηση. Κρατά και τα δύο κομμάτια στο, στο σκάφος και αυτό θεωρείται ως επεξεργασία. Η παρούσα νομοθεσία κατ' εξαίρεση επιτρέπει κάποια σκάφη και στο πλήρωμα να αφαιρούν τα πτερίγια με την προπόθεση ότι διατηρούν το σώμα ε, επί του σκάφου και διάφορου άλλου όρου εν πάση περιπτώσει, που δεν χρειάζεται να σα πω λεπτομερώς, αλλά εν περιπτώσει θα πρέπει να τονίσω ότι η αφαίρεση των πτερυγίων και η απόρριψη του σώματο ήδη απαγορεύεται, απλώ υπάρχει αυτό το παραθυράκι που σε ορισμένε περιπτώσεις επιτρέπει την αφαίρεση των πτερυγίων όπου και να περάσει αυτό χωρί να εντοπιστεί, γιατί αυτό είναι ένα από τα κύρια προβλήματα και του λόγου του οποίου οφείλεται η τροποποίηση του κανονισμού θέλουμε να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να ανοιχνεύσουμε οποιαδήποτε πράξη αφαίρεση πτερυγίων. Τώρα, θα προσπαθήσω με την αντίστροφη σειρά να απαντήσω στη τελευταία ερώτηση, δηλαδή αν βλέπουμε καμιά, κάνα παραθυράκι, αν κάποιος νομοθέτης στην Επιτροπή έχει, κάνει, έχει βρει κάποιο παραθυράκι. Εγώ είμαι λόγος θαλάσσιος βιολόγος, δεν είμαι νομικός. Έχω φυσικά έρθει σε επαφή με τους ε, νομικούς μας. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει εδώ παραθυράκι και κανείς δεν μου έχει υποδείξει εδώ παραθυράκι. Αν το πτερίγιο είναι πάνω στο σώμα του καρχαρία και οι επιθεωρητές δουν ότι τα πτερίγια όλα είναι πάνω στο σώμα του καρχαρία, ε, δεν θα μπορεί να υπάρξει παραθυράκι. Είναι προφανές για έναν επιθεωρητή. Έχω ίσως λίγο καιρό και σύντομα θα προσπαθήσω να απαντήσω σε άλλα σχόλια. Αυτό που προτείνουμε και θέλω να το υπογραμμίσω δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε εξαίρεση σε αυτήν την πρόταση δεν προβλέπουμε καμιά εξαίρεση. Όλοι οι καρχαρίες θα πρέπει να εκφορτώνονται με τα πτερήγια τους πάνω τους, φυσικά ε, συνδεδεμένα. Και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την αποθήκευση, την ασφάλεια, την ποιότητα κτλ. Πιστεύουμε πως αυτή η τεχνική λύση και άλλες λύσεις που έχουμε προτείνει στο πλουστάσιο μας θα καλύψουν όλους τους, όλες τις ανησυχίες του τομέα που μας ενημέρωσε και τις ανησυχίες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αυτά είχα να σας πω γιατί τελείωσε και ο χρόνος μου. Σας ε, ζητώ συγγνώμη, ε, ε, αλλά έχουμε άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι επίσης σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω που σε τόσο σύντομο χρόνο μπορέσατε να μας δώσετε και τον ορισμό και μας απαντήσατε και στο ερώτημα. Ο εισηγητής θα ήθελε πάρει το λόγο, κύριε Τσανώνη. Δύο λεπτά. Νομίζω πως όλα τα ζητήματα έχουν διευκρινιστεί, δεν υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες, οπότε το μόνο που μπορούμε να πούμε να ευχηθούμε να εγκριθεί όταν θα πάει για ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζανώνη. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 7 Μαρτίου στις 12 η ώρα. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θα ψηφιστεί 25-26 Απριλίου ε, και στην Επιτροπή Αλίας που είναι αρμόδια επί της ουσίας, στις 30 Μαΐου. Στην Ολομέλεια του Ιουλίου θα ψηφιστεί η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ε, σύντομες και περιεκτικές παρεμβάσεις σας είναι σημαντικό θέμα Είναι σημαντικό να σταματήσει η πρακτική αυτή και να έχουμε σαφείς ε, κανόνες. Προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης ε, που είναι το σημείο 8. Ε, το θέμα εδώ είναι η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του Κιώτο. Οι συντονιστές αποφάσισαν τον Οκτώβριο να καλέσουμε έναν εκπρόσωπο της Κομισιόν για να συζητήσουμε και να ακούσουμε σε τι βαθμό ε, ε, πληρούνται οι στόχοι του Κιώτο. Η Ναταλή Φεστέη έχει το λόγο εκ μέρους της Κομισιόν. Παρακαλώ, δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Thank you um, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εσάς και την ε, Επιτροπή σας που καλέσατε την Κομισιόν και της δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσματα της έκθεσης της ε, σχετικά με την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων του Κιώτο. Όπως ε, ξέρετε η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, είναι συνυπεύθυνα για την ε, μείωση των ε, εκπομπών και κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιώτο στη Νέα το 1999 η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι εκείνη και τα κράτη-μέλη θα πληρώσουν από κοινού του, τις προϋποθέσεις του πρωτοκόλλου του Κιώτο. Δεδομένων λοιπόν ε, των ε, σχετικών απαιτήσεων ε, για έλεγχο των εκπομπών, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της πολιτικής για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να αναλύονται σε τακτική βάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συντονίζει τις προσπάθειες ε, που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφωθεί με το πρωτοκόλλο του Κιώτο. Από την αρχή της θέσης ισχύ του πρωτοκόλλου ε, του Κιώτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τους στόχους. Ε, αναφέρομαι στο έγγραφο 624 ε, μαζί με το ε, έγγραφο των υπηρεσιών της Κομισιόν. Να σας θυμίσω αρχικά τις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν, σύμφωνα με την UNFCCC και την ΚΕΙΠΗ, τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν έπρεπε να μειώσουν κατά 8% ε, τις ε, εκπομπές τους ε, σε σχέση με, την, με το έτος αναφοράς και τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 έχουν στόχους για μείωση από 6 έως 8%. Η Μάλτα και η Κύπρος δεν έχουν τέτοιες υποχρεώσεις. Επίσης υπάρχουν οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώριο επίπεδο, δηλαδή η μείωση ε, εκπομπών ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα κατά 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 1990. Ε, όσον αφορά τις εκπομπές έχουμε την εξή εικόνα. Για ε, τα 27 κράτη-μέλη βλέπουμε μείωση 15,5% σε σχέση με το 1990. Ε, και για τα 15 κράτη-μέλη βλέπουμε μείωση 10,7% σε σχέση με το έτος αναφοράς και το 2010. Αν αναλύσουμε ανατομέα το μερίδιο, ε, των εκπομπών βλέπουμε ότι, και μας το δείχνει αυτό η έκθεση, ότι η παροχή ενέργειας ε, προσωπεύει το 31,8%, ε, οι μεταφορές 19,7%, η βιομηχανία 7,3%, η γεωργία 9,9%, τα απορρίμματα 3%, οι διαλύτες και άλλα 0,2%. Η έκθεση προόδου δείχνει επίσης και σας παραπέμπω ε, στο διάγραμμα το οποίο ε, ε, είναι αυτονόητο ότι εάν συνεχίζαμε όπως πριν θα είχαμε συνεχή αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ενώ η γραμμή που ακολουθούν τα 15 πρώτα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μα δείχνει ότι έχουμε φτάσει κάτω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιώτο. Επίσης βλέπουμε ότι όπως δείχνει η ετήσια έκθεση πρόοδου μας, ε, ότι είχαμε αύξηση των εκπομπών ε, στο διάστημα 2009 με 2010. Βλέπουμε όμως ότι και με τα υπάρχοντα μέτρα θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε σε τάση μείωσης και με περαιτέρω μέτρα μείωση ε, θα ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω η πτωτική αυτή τάση. Στις 7 Οκτωβρίου πέρσι η Κομισιόν υιοθέτησε την ετήσια έκθεσή της και το βασικό μήνυμα είναι ότι πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παραμένει καθοδόνη για την επίτευξη των ε, στόχων ε, του και όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παρά την αύξηση 2,4% των εκπομπών το 2010. Η αύξηση αυτή ακολουθεί μετά από πτώση 7% το 2009 που σε μεγάλο μέρος οφειλόταν στην η οικονομική ύφεση και στις βιώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, με πολιτικές δράσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καταφέρνει να αποσυνδέσει τις εκπομπές από την ε, αύξηση του ΑΕΠ. 15,5% έπεσαν οι εκπομπές ανάμεσα στο 1990 και ε, στο 2010, ενώ η οικονομία αυξήθηκε κατά ε, περίπου 40%. Ε, ε, είδαμε ότι η πτώση για το... οι στόχοι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιώτο, θα ξεπεραστούν και ε, τα μέτρα προβλέπονται να οδηγήσουν σε μείωση 10,5% σε σχέση με ε, το έτος αναφοράς. Η αγορά των ε, ποσοστώσεων από τρίτες χώρες θα οδηγήσουν περαιτέρω σε μείωση. Επιπλέον 10 από τα 12 κράτη-μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 και που έχουν υποχρέωση μείωση ε, βρίσκονται επίση καθοδόν ε, ω προ την μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Γενικά λοιπόν είναι σχετικά αισιόδοξη η έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να πληρώσει τον στόχο τη ε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιώτο παρά την αύξηση πέρσι καθότι οι εκπομπές ε, τη ευρωπαϊκή Ένωση ήδη βρίσκονται 10,7% κάτω από το έτος αναφοράς. Επιπλέον ε, φαίνεται ότι ε, ότι οι εκπομπές από το 2008 μέχρι το 2012 θα είναι 10,5 κάτω από το έτος αναφοράς ε, και ότι η συνολική μείωση μπορεί να φτάνει το 13,4% αν όλα τα μέτρα όπως η χρήση των κυβερνήσεων ε, του μέσου για το διοξείδιο του άνθρακα ε, επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λοιπόν ε, βρίσκονται καθοδόν και μόνο τρία κράτη-μέλη, η Αυστρία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο, ίσως ε, αντιμετωπίσουν ε, δυσκολίες ε, στην επίτευξη των στόχων χωρίς να υπονομεύουν όμως την δυνατότητα των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής, τότε κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να πετύχουν τους στόχους τους. Η Φιλανδία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται καθοδόν να πετύχουν τον εγχώριο στόχο τους και ε, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο ευελιξίας του Κιώτο, Μόνο τρία κράτη-μέλη, η Αυστρία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων τους χωρίς όμως αυτό να υπονομεύει τη δυνατότητα των 15 κρατών ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχουν τους στόχους τους. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό ότι όπως είπα και πριν, ε, στα περισσότερα από τα 12 κράτη-μέλη που ε, προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, είδαμε μια ελαφρά αύξηση από το 2008 και το 2009, αλλά εννέα από αυτά που έχουν στόχο ε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιώτο αναμένεται να τον πετύχουν ή να τον ξεπεράσουν κιόλα. Έχουμε λοιπόν ε, το, τον μηχανισμό ευελιξίας ε, του Κιώτο. η Κύπρος και η Μάλτα δεν έχουν υποχρέωση μείωση των εκπομπών τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιώτο. Όπως είπα στην αρχή της παρουσίασης αυτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει δεσμευτεί μέχρι το 2020 ε, σε εγχώριο επίπεδο να μειώσει εκπομπές, ε, έτσι ε, κοιτώντας πέρα από τους στόχους του Κιώτο. Αυτός ο εγχώριος στόχος προβλέπει μέχρι το 2020 να μειωθούν οι εκπομπές να μειωθούν κατά το 20% σε σχέση με το 1990. Στη ε, έχει συμπεριληφθεί στην ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020 ε, ο στόχος αυτός και η και ο στόχος μείωσης των εκπομπών είναι ένας από τους πέντε βασικούς στόχους. Σε σχέση με το 1990, μιλάμε για μείωση κατά 14%. Μείωση μείον 1% σε σχέση ε, με το 2005. Και έχουν οριστεί ε, διάφοροι στόχοι μέχρι το 2020. Όσον αφορά τον εγχώριο αυτών στόχων, η έκθεση δείχνει την ε, υπολογισμένη επίτευξη των στόχων και καταλήγει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να πετύχουν τους στόχους τους με τις πολιτικές που ήδη υπάρχουν. Επιπλέον, 7 κράτη-μέλη θα πετύχουν τους στόχους όταν ε, ληφθούν πρόσθετα μέτρα και πολιτικές ε, τα οποία θα επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ενώ τα υπόλοιπα 9 κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν πρόσθετες πολιτικές για να πετύχουν τους στόχους τους. Στην πράξη λοιπόν, ε, αν κοιτάξουμε τους ε, στόχους ε, για το 2020. Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες ιδιαίτερα στον τομέα των οικοδομών, των μεταφορών, της γεωργίας και των απορριμμάτων. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει τα πρόσθετα αυτά μέτρα για να επιτύχουν το στόχο του 2020 και μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε ε, πολύ πιο ε, σημαντικές μειώσεις των εκπομπών. Γενικά, το μήνυμα της έκθεσης αυτής είναι ότι ε, η αύξηση κατά 2,4% στις εκπομπές μπορεί να εξηγηθεί με την ανάπτυξη που είδαμε, την οικονομική ανάπτυξη, ανάκαμψη που είδαμε σε κάποιες χώρες. Ε, επίσης, ο, ο ιδιαίτερα κρύος χειμώνας ε, αύξησε την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. Ταυτόχρονα η έκθεση δείχνει ότι η αύξηση των εκπομπών περιορίστηκε από μεταφορά προς το φυσικό αέριο από τον ε, άνθρακα ως καύσιμο. Ε, οι διαφορετικές αλλαγές λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν θετικές επιπτώσεις. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που μας επιτρέπει έκθεση να τονίσουμε είναι ότι βλέπουμε συνέχιση της αποσύνδεσης ε, των εκπομπών από τον ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Και είδαμε για παράδειγμα μείωση κατά 7% των ε, εκπομπών ενώ ε, η συρρήκνωση της οικονομίας ήταν πολύ χαμηλότερη. Θέλουμε λοιπόν, ε, βλέπουμε λοιπόν ότι οι προσπάθειές μας να ε, γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινωνία χαμηλών εκπομπών ε, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και χρειάζονται κάποιες επιπλέον προσπάθειες για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank, Frau Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική παρουσίασή σας. Ε, σχετικά με την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων του Κιώτο. Ε, αναφερθήκατε στα 15 πρώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω εδώ κατάλογο των ομιλητών. Πρώτα ο Μάρτιν Κέλενεν και κατόπιν ε, η Φιουζέ. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαστε υπέρ τη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικώ, αλλά προτιμούμε τον ρεαλισμό παρά την ρητορική δυνότητα. Μόνο έτσι θα υλοποιήσουμε του στόχου, γιατί υπάρχει ε, κίνδυνος να χαθούμε στου ευθέρωτους ε, θεωρητικούς στόχους, ε, αντί να λάβουμε συγκεκριμένε ε, συλλογικές δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Η έκθεση δείχνει ότι κάποια κράτη-μέλη ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίε προκειμένου να διατηρήσουν την αρχική του πρόοδο ως προς την υλοποίηση των στόχων. Και αναφυσβήτητα η οικονομική κρίση αποδυνάμωσε την πολιτική βούληση και την αίσθηση του κατεπήγοντος για την υλοποίηση των στόχων σε πολλές χώρες. Μέσω της κρίση, λοιπόν δεν έχουμε την πολυτέλεια για περαιτέρω μονόπλευρες ε, αναλήψεις δεσμεύσεων εις βάρος της ανταγωνιστικότητας ε, της βιομηχανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε αντίστοιχες προσπάθειες και από άλλες εκβιομηχανισμένες χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά και ε, λογικές και δίκες ε, ε, δεσμεύσεις και από αναδυόμενες οικονομίες και αναπτυσσόμενες χώρες. Στο μέλλον θέλουμε περισσότερη αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων και η οικονομική ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ίσως να προωθηθεί με μια βιομηχανία που θα είναι πιο αποδοτική ενεργειακά αλλά και από κυβερνήσεις που θα προσαρμόζουν τους ενεργειακούς στόχους ε, στις ε, περιστάσεις, ε, αλλά δεν θα χάνουν την ευρύτερη προοπτική. Κάτι άλλο που με απασχολεί εδώ και καιρό. Έχετε κάνει κάποιες προβλέψεις, γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχω ακούσει, για το κατά πόσο έχει λάβει η χώρα κάποια μείωση στις εκπομπές για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλες που έμεσα παράγονται. Για παράδειγμα, στις διάφορες πολιτικές, στις κοινοτικές, τι μείωση διοξιδίων του άνθρακα ε, έχουμε ή τι, ε, με τις μετεγκαταστάσεις των μηχανιών, τι τμήμα τους έχει ε, μεταφερθεί ουσιαστικά σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιφκοσέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ Συνεχίζοντα τον προβληματισμό και τι ερωτήσει του προλαλήσαντο, ήθελα και εγώ να θέσω τρει ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερώτηση πρώτη. Τι προβλέψει για τι μειώσει που μα ε, περιγράφει στην έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι οφείλεται στο φαινόμενο της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Μήπω ε, η μείωση των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε ένα είδους ε, αποβιομηχανοποίηση τη Ευρωπαϊκής Ένωση λόγω της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων. Ναι, μεν έτσι έχουμε μείωση των ε, εκπομπών καυσαερίων, αλλά έχουμε ολέθρια αποτελέσματα στις βιομηχανίες μας. Ποιο τμήμα λοιπόν της μείωσης οφείλεται στη μετεγκατάσταση των εργοστασίων από το 1990 και μετά. Και η λογική απόρρια της παρατήρησης αυτής είναι, και της ερώτησης είναι μήπως θα πρέπει να θεωρούμε ως ευρωπαϊκές εκπομπές τις φές αυτές εκπομπές ή την ε, φαιά αυτή ενέργεια που περιλαμβάνεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που εμείς εισάγουμε από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εδώ καταναλώνουμε αυτά τα προϊόντα. Γιατί για, την, για τις εκπομπές μιλούμε μόνο για την παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφορές, βιομηχανία, οικοδομές και το καθεξής. Αλλά έχουμε και την κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισάγουμε πολλά προϊόντα που περιέχουν από το λόγο από τον τρόπο παρασκευής τους τις εκπομπές, παρόλο που δεν έχουν γίνει αυτές οι εκπομπές, δεν έχουν εκλειθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ό,τι αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών, πρόκειται για το μηχανισμό και το Κιώτο, είναι ένας μηχανισμός ελαστικότητας. Μήπως όπως υπάρχουν παρεκτροπές έως και καταχρήση και διαφθορά στη χρήση αυτού του τρόπου εμπορίας εκπομπών και σε αυτή την αγορά των εκπομπών των καυσαερίων. Μήπως θα μπορούσε να μας ενημερώσει πιο διεξοδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τελευταία παρατήρηση. Φαίνεται ότι η επιστήμη, και εδώ μιλώ για τους φίλους επιστήμονες της ΖΕΚ που φαίνεται ότι λένε σε σχέση με την πρώτη έκθεσή τους πριν από μία εικοσαετία και σε σχέση με την τελευταία πριν από μία ετία αναμένεται και νέα επιστημονική έκθεση το 2014 και γνωρίζουμε από τις εκθέσεις αυτές ότι ε, τα καυσαέρια και τα αποτελέσματα των καυσαέριων δεν είναι γραμμικά. Μπορεί να έχουμε ένα είδος ε, θετικής ε, ε, αναδρομικής ισχύω, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις του μεθανίου ε, που μπορούν να περάσουν ε, και να οδηγήσουν σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Περιμένουμε σε δύο χρόνια την επιστημονική έρευνα, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι στόχοι δεν είναι μόνο γραμμικοί. Μερικές φορές υπάρχουν και τα κατόφλια και πολλές φορές κάποια θετική αναδρομική δράση για, την, για το λιώσιμο των πάγων για παράδειγμα και για την απότομη έκκληση μεθανίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι στις δύο ερωτήσεις που έγιναν εδώ πέρα. Όταν θέτουμε στόχους στην Ευρώπη, ότι η Ευρώπη ε, θα πρέπει να ε, μειώσει κατά 30-40%, ε, Βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντική η βούληση. Όταν όμως μιλάμε για συγκεκριμένα μέτρα, τότε είναι περιορισμένη η βούληση, διότι φοβόμαστε ότι αυτό θα οδηγήσει σε μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων. μπορείτε να έχετε αποτελέσματα σχετικά με τις συνέπειες της ε, οικονομικής ε, κρίσης ε, και τι γίνεται με τις επενδύσεις στην Ευρώπη και τις επενδύσεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Έχετε σχετικά δεδομένα, διότι νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα σε όλη την νομοθεσία που έχει να κάνει με την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος τι σημαίνουν ε, όλα αυτά για την οικονομική ανάπτυξη, διότι το κλίμα δεν το νοιάζει ε, αν ε, γίνονται οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλα μέρη του κόσμου. Θα σας παρακαλούσα συγκεκριμένη απάντηση αν έχετε τέτοιες... θα, παρακαλούσα πολύ να μου δώσετε τέτοια στοιχεία αν υπάρχουν. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Thanks a lot. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις. Επανειλημμένως ε, εκφράστηκε η ανησυχία για το πεδίο των ε, δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την ε, έκθεση και τη δυναμική του βιομηχανικού κλάδου σε σχέση με τις οικονομικές αντικσότητες και τις δυσκολίες ε, που δημιουργούν σε απώλεια ανταγωνιστικότητας οι στόχοι αυτοί. Και επίσης ε, υπάρχει και η τάση να βοηθήσουμε εντό εισαγωγικών τη μείωση ε, των καυσαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μετεγκατάστασης των εργοστασίων και των επιχειρήσεων, δηλαδή ουσιαστικά από μια αποβιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει που είναι οι μετρήσεις ε, των εκπομ... της μη... η ε, μετρήση των μείωσης εκπομπών καυσαερίου στην Ένωση μήπως ε, δίνει αποτελέσμα... δίνουν αποτελέσματα που οφείλονται στη μετεγκατάσταση σε μεγάλο βαθμό για παράδειγμα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η έκθεσή μας χρησιμοποιεί στοιχεία των κρατών μελών, τα συγκεντρώνει, τα αναλύει και κατόπιν τα θέτει υπό μια πολιτική και στατιστική προοπτική. Η στατιστική προοπτική οδηγεί στα στοιχεία που σας παρουσίασα εδώ. Η πολιτική προοπτική εξηγείται και από την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πέρυσι το Μάρτιο υιοθέτησε το δικό χάρτη για την Ευρώπη μέχρι το 2050 που λέει ότι από τη στιγμή που θέλουμε σφαιρική δράση και όχι κατακαιρματισμένη, θα υλοποιήσουμε το στόχο της μείωσης κατά 2 βαθμού Κελσίου μέχρι το 2050. Και κατακαιρματισμένη δυστυχώ είναι η δική μας ικανότητα που περιορίζεται σε 14% των παγκοσμίων εκπομπών. Οπότε ναι, μεν σε στατιστικό επίπεδο η έκθεση παρουσιάζει τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη τις δυναμικές εξελίξεις εξαιτία των αποφάσεων των επιχειρήσεων για μετεγκατάσταση, μετατόπιση των δραστηριοτήτων, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η μείωση των εκπομπών, η ανάγκη της μείωσης ε, είναι όχι να, όχι να ενισχύσει τη μετεκατάσταση. Και υπάρχει και η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να πει ότι η παγκόσμια στόχοι, δηλαδή η μείωση της θερμοκρασίας μέχρι το 2050, θα πρέπει ε, να γίνονται με σφαιρικό και όχι κατακαιρματισμένο τρόπο. Αυτά θα ήθελα να πω προς το παρόν. Um, ε, σε ό,τι αφορά την ε, ερώτηση για την ε, κατά πόσο η προσέγγιση μας βασίζεται στην παραγωγή. Ναι, αυτό κάνουμε τώρα. Ξεκινάμε με κάποιες συζητήσεις για μια προσέγγιση που θα εστιάζεται στην κατανάλωση, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολη την προσέγγιση που εστιάζεται στην παραγωγή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι η μόνη, το μόνο όργανο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα θέματα αυτά και με όλα τα συναφή ζητήματα που ε, οφείλονται σε μια προσέγγιση που θα εστιάζεται στην κατανάλωση. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο think tank που αντιμετωπίζει ακριβώς τις ίδιες δυσκολίες προσπαθώντας απελπισμένα να ε, υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα στηρίζεται στην αλυσίδα ανεφοδιασμού. Και σε μια μελέτη της αλυσίδας ανεφοδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη περισσότερο την κατανάλωση από ό,τι την παράγωγη. Πάντως δεν είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο και ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για να υιοθετήσουμε μια τέτοια προσέγγιση που θεστιάζεται στην κατανάλωση. Πάντως, όντω μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα και μας απασχολεί. Αναφερθήκατε και στην αναμενόμενη έκθεση GEC για το 2014, την επιστημονική μελέτη στην πολιτική μας και στην έκθεση μας αυτή λαμβάνουμε υπόψη τα επιστημονικά πορίσματα. Οι εκθέσεις μας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαμβάνουμε υπόψη τα επιστημονικά πορίσματα στις δικές μας εκθέσεις. Τώρα, οι εξελίξει της μειώση εκπομπών δεν είναι γραμμικές. Το γνωρίζουμε αυτό, συμφωνούμε. Έχουμε πολύ ρεαλιστική προσέγγιση και προσπαθούμε να αντιληφθούμε αυτή την έλλειψη γραμμικότητας σε ορισμένε περιπτώσεις. Δεν έχουμε μια προ... προκαθορισμένη, προκατηλημένη αντίδραση και όταν οι γραφικές παραστάσεις δίνουν γραμμική εξέλιξη, δίνουν το μήνυμα απλώς ότι η προσέγγιση είναι ε, σαν να μην συνέβαινε τίποτα διαφορετικό και οπότε μια τέτοια γραμμική εξέλιξη μας βγάζει από το πεδίο μας. Σε ό,τι αφορά την ελαστικότητα του συστήματος εμπορίας εκπομπών και τις παρεκτροπές ή τη διαφθορά που παρατηρείται μερικές φορές στην αγορά. Το γνωρίζουμε, αλλά εμείς λάβαμε όλα τα δυνατά μέτρα για να εξασφαλίσουμε διαφάνεια του συστήματος εμπορίας εκπομπών και φυσικά πήραμε και όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να βρίσκεται υπό έλεγχο η κατάσταση και οποιαδήποτε, οποιασδήποτε παρεκτροπές να διορθώνονται άμεσα. Δεν νομίζω ότι αυτές οι εξαιρέσεις, αυτά τα επεισόδια είναι ε, ε, ο κανόνας. Νομίζω ότι υπάρχει διαφάνεια και μεγάλη εντιμότητα γενικώ στην εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική σας απάντηση και την ε, πολύ καλή ε, παρουσίασή σας. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Ακούσαμε και τις ε, απόψεις των συναδέρφων από δύο πολιτικές ομάδες. Πιστεύω ότι χρειάζεται εδώ, χρειάζεται εδώ πέρα μια περισσότερο εις βάθος ανάλυση, διότι νομίζω ότι η συμφωνία ή όχι με ε, μελλοντικά νομοθετήματα συνδέεται πάρα πολύ στενά με το θέμα αυτό. Είναι λοιπόν, ε, και επειδή ο φόβος ε, δεν είναι καλός σύμβουλος, είναι πολύ καλό να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό για να δείξουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να αποσυνδεθεί από το θέμα των ε, εκπομπών. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, χρειαζόμαστε όμως ε, περισσότερες εξηγήσει και περαιτέρω ανάλυση. Διακόπτω εδώ την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και σας παρακαλώ στις 3 η ώρα να είσαστε παρόντες διότι θα ξεκινήσουμε με τις ε, ψηφοφορίες. Να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας σας και σας εύχομαι ε, καλό μεσημέρι.